Ε, ladies Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίε και κύριοι, να ζητήσω συγγνώμη για την ελαφρά καθυστέρηση. Αλλά διεξάγεται μια διάσκεψη στο Κοινοβούλιο με πολλούς εκπροσώπους ε, και άργησε κάπου να ξεκινήσει. Χρειάστηκε να κάνω την αναπτήρια ομιλία εγώ. Είναι η πρώτη μας κοινή συνεδρίαση των δύο επιτροπών μας και χαίρομαι ιδιαίτερα. Κυρία Πρόεδρε, χαίρομαι που μπορούμε να συμπροεδρεύσουμε τόσο στην σημερινή συνεδρίαση όσο και στην προσεχή. Αν δεν υπάρχουν σχόλια σχετικά με μέσα διάταξη, μπορούμε να την εγκρίνουμε. Δεν βλέπω να υπάρχει κάποιος που να ζητάει το λόγο. Η διερμηνία παρέχεται σε όλες τις γλώσσες της Ένωσης εκτός των Μαλτέζικων, Κροατικών και Σλοβενικών. Ενημέρωση σχετικά με διαδικασία. Είναι πολύ σημαντικό ζήτημα. Συντάξαμε από κοινού σημαντικές εκθέσεις. Θα ήθελα να συγχαρώ πρώτα απ' όλα όλους ε, όσοι ενεπλάκησαν στην διοργάνωση και στην σύνταξη ε, αυτών των εκθέσεων για την πολύ καλή συνεργασία και την εξαιρετική εργασία που έγινε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την κυρία Φόρουσα για τις δραστηριότητές της αλλά και τους δύο συνεισηγητές, την κυρία Γκέπχαρτ και η κυρία Κάλλας. Η έκθεσή μας θα συζητηθεί και θα εγκριθεί σε κοινή συνεδριάσει των δύο επιτροπών μας. Θα υπάρξει και μια χωριστή ημιστεδιάρξη για κάθε συνάντηση υπό την κοινή προεδρία των δύο προέδρων. Έτσι αποφασίσαμε νομίζουμε ότι είναι η καλύτερη λύση αυτή το σχετικά με τη διαδικασία μας, αν υπάρχουν ερωτήσεις ή σχόλια, περνάμε στο σημείο 3 της μεσαίας διατάξεως προς ε, μια πράξη ενιαία ψηφιακής αγοράς. Κυρία Συμπρόεδρε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια και ευχαριστώ και τους ε, συμμετέχοντες ε, στην αίθουσα. Στο βάθος βλέπω ότι υπάρχουν και στα θεωρία πολύ οι οποίοι δείχνουν ότι η, ψηφιακή αγορά τους ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Ο κ. Μπούζεκ ε, θα προεδρεύσει τον πρώτο γύρο της ε, σημερινής συνεδρίας κατά τη συζήτηση των σκιωδών και των εισηγητών και εγώ θα προεδρεύσω στο δεύτερο γύρο όπου Όσοι επιθυμούν να λάβουν το λόγο μπορούν να το ζητήσουν από τώρα διότι έχουμε αρχίσει να συντάσσουμε τον κατάλογο των αγοριτών. Σιγά σιγά, μην βιάζεστε. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να καταγράψουμε τα ονόματά σας ε, προοδευτικά. Κρατήστε το καρταλάκι αναρτημένο μέχρι ότου να σας ε, ενημερώσουμε. Έχουμε τους συντονιστές ε, στον πρώτη σειρά και τους αντιπροέδρους ε, και τους κοιόδες εισηγητές στην δεύτερη σειρά των εδράνων. Πρέπει να παραμείνουμε εντός χρονικών ορίων και στην αρχή της δεύτερης ε, συνεδρίας θα αναγνώσω τον κατάλογο των αγορητών έτσι ώστε αν δεν έχει ε, συμπεριληφθεί κάποιο όνομα, μπορείτε να μας ενημερώσετε. Ευχαριστώ πολύ, συνεχίζει ο κύριος Μπούζεκ. Να πω προς τους προσεγγλημένους, προς τους επισκέπτους, ότι οι επιτροπές μας, σε επιτροπές μας συμμετέχουν περίπου 120 μέλη, ...751 συνολικά τα μέλη του Κοινοβουλίου στις κοινέ μας συνεδριάσεις στο Κοινοβούλιο και τις ψηφοφορίες. Αυτή η αίθουσα στην οποία βρισκόμαστε σήμερα είναι γεμάτη πλήρης βουλευτών. Έχουμε και τους βοηθούς μας, τους συμβούλους, πολιτικούς συμβούλους που παρευρίσκονται σε αυτήν την αίθουσα αλλά στις στην έδρανα συμμετέχουν ε, τα μέλη των δύο επιτροπών, περίπου 120. Αυτά για να γνωρίζουν οι επισκέπτες μας. Μπορείτε φυσικά να ακούσετε όλες τις γλώσσες σχεδόν. Σήμερα 21 γλώσσες της Ένωσης είναι στη διάθεση σας. Πέραμε λοιπόν στην ε, έκθεση. Όπως γνωρίζετε, η στρατηγική για την ενία αγορά εγκρίθηκε από την ε, Κομισιόν τον, ε, τον Μάιο του 2015 και τώρα έχουμε ενώπιόν μας την πρόταση της Κομισιόν με 16 δράσεις κλειδί κλειδιά συγγνώμη και θέλουμε να τις ελέγξουμε και να προτείνουμε τις ε, θέσεις μας διότι όλοι θα πρέπει να ολοκληρωθούν το 2016. Έχει μεγάλη σημασία λοιπόν να προτείνουμε κάτι το αυτό, το συγκεκριμένο. Καλύτερη πρόσβαση στα ψηφιακά αγαθά. Αυτό είναι ο βασικό στόχο των συζητήσεών να δημιουργήσουν τι καλύτερε προποθέσει, ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού και δυναμικό ε, αύξηση και ενίσχυση της ψηφιακής ε, αγοράς θα ζητήσουμε από τους συζητητές μας ε, και από τους δύο να μας παρουσιάσουν τις εκθέσεις τους 7 λεπτά έκαστος και επίτα οι σκιώδεις συζητητές ή τους ε, αναπληρωτές τους να λάβουν το λόγο για 3 λεπτά έκαστος και αργότερα όλοι οι υπόλοιποι συνάδελφοι όπως είπε και η συμπρόεδρος νωρίτερα. Αρχίζουμε λοιπόν με τους συζητητές με σειρά η κυρία Εύελη Γκέπχαρντ, πρώτη ομιλήτρια και μετά η κυρία Κάλλας. Εύελη, έχει το λόγο. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα αυτή σε αυτόν τον χώρο να διαμορφωθεί αυτή η συνεδρίαση. Και προτού υπησέθω στο θέμα, θα ήθελα ιδιαίτερα την συνεισηγήτρια κυρία Κάλλας να την ευχαριστήσω για μια πραγματικά πολύ επικοδομητική συνεργασία και στους τομείς εκείνους επί των οποίων δεν είμαστε της ίδιας γνώμης και δεν συνενούσαμε. Καταφέραμε να καταλήξουμε σε σωστές αποφάσεις και αυτό είναι κάτι καλό. Και υστερότερα θα αναφερθώ σε αυτές τις διαφωνίες, διότι πρέπει να συζητηθούν αυτά τα θέματα φυσικά. Διότι δύο εισηγήτριες δεν αντανακλούν τις απόψεις τους απλώς, αλλά την άποψη 751 ευρωβουλευτών και με βάση μια καλή συζήτηση μπορούμε να λάβουμε μια τέτοια κοινή απόφαση. Είναι ειδική πρόκληση με αυτό το άρθρο 55 <clears throat> που ε, δεν ήθιστε στο κοινοβούλιο μας και στο, με το άρθρο 54 με την, ε, τις συνεμπλεκόμενες επιτροπές ε, και τις εκθέσεις και με το άρθρο 53 επιπρόσθετα να προχωρήσουμε. Προσδοκώ να δω πώς θα προχωρήσουν οι εργασίες αυτές και τι θα γίνει τελικά, ποια έκβαση θα έχουμε διοργανωτικά καταφέραμε να πετύχουμε αρκετά πράγματα και έτσι αυτή η καλή εργασία είναι θετικό γεγονός και εργαζόμαστε θετικά. Αυτό το θέμα και αυτό δείχνει και την απήχηση στο Ευρωκοινοβούλιο αλλά και εκτός Ευρωκοινοβουλίου αυτό το θέμα είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό θέμα διότι βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή μέσα στον πυρήνα μιας επανάστασης, μιας ψηφιακής επανάστασης που σε όλους τους τομείς της ζωής και εργασίας, σε όλους τους τομείς της κοινωνίας ε, προχωρεί. Και αυτό τι σημαίνει, ότι σε αυτά τα θέματα φυσικά ευρύτατα θα πρέπει να τοποθετηθούμε και να βρούμε αποφάσεις, να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις και πέρα από τις προκλήσεις αυτές. Προκλήσεις που ολιστικά, σφαιρικά πρέπει να αντιμετωπιστούν, διότι όχι μόνο σε επιμέρους σημεία <clears throat> μπορούμε τα αποτελέσματα να τα εξετάσουμε, αλλά συνολικά στο σύνολο των αποφάσεων που πρόκειται να λάβουμε και θα ληφθούν και να δούμε τι θα γίνει τελικά. Αυτές τις αλλαγές τις βρίσκουμε και στον κόσμο της βιομηχανίας και των εργοστασίων και των παραγωγών. Έχουμε μια νέα πραγματικότητα, νέα πράγματα μπορούν να δημιουργηθούν που πριν από τρία-τέσσερα χρόνια δεν τολμούσε κανείς να ονειρευτεί ότι θα μπορούσε να γινόταν. Και έχουμε και καινοτομικά, καινοτόμα έργα σε αυτόν τον τομέα. Υπάρχουν πολλά σημεία και όσον αφορά τις υπηρεσίες, με πλατφόρμες, με την sharing economy, την ε, επιμεριζόμενη οικονομία κοινών δράσεων και που μας θέτουν προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Και φυσικά υπάρχουν και πολλές αλλαγές, μεταβολές, και εξελίξει σε αυτούς τους τομείς. Πώς θα συνεργαστούμε και θα εργαστούμε στο μέλλον σε αυτόν τον νέο κόσμο εντός εισαγωγικών. Τι θα γίνει με την ε, διαχείριση και την διακυβέρνηση. Τι θα κάνουν τα κράτη με όλα αυτά. Και έχουμε φυσικά και ε, νέους τομείς ε, ηλεκτρονικών δραστηριοτήτων και όλα αυτά προϋποθέτουν ότι εμείς καταρχήν θα προσέξουμε πολύ προσεκτικά ποια συνέχεια θα δώσουμε. Τι βρίσκεται στο τραπέζι ως προτάσεις. Πώς θα τα αναλύσουμε όλα αυτά. Να δούμε ποια επιτεύγματα μπορούν να απορρέουν από όλα αυτά ποιες είναι οι προκλήσεις αλλά που βρίσκονται και οι κίνδυνοι και που βρίσκονται ανάγκες και αναγκαιότητες που νομοθετικά θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Όλα αυτά είναι θέματα που σήμερα δεν έχουμε έτοιμες απαντήσεις. Δεν μπορούμε να πούμε ότι πρέπει όλα αυτά να γίνουν με τον ένα ή άλλο τρόπο. Πρέπει να δούμε, να σκεφτούμε πρώτα τι είναι αναγκαίο και τι όχι. Το πρώτο θέμα που πρέπει να εξετάσουμε σε αυτόν τον τομέα είναι τι θα κάνουμε με τις υποδομές. Δηλαδή πώς θα λειτουργήσουν όλα αυτά. Και την Πέμπτη, για παράδειγμα, είχα μια συζήτηση με Γεωργού την προηγούμενη Πέμπτη. Μας λένε, είναι τεράστια πρόκληση αυτή. Μας απαιτεί, από εμά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις πληροφορίες μας, εμείς, ψηφιακά να τις διαβιβάζουμε. Αλλά σε κάποιους τομείς, σε κάποια μέρη αυτής της χώρας δεν έχουμε τέτοια κάλυψη Πρέπει με μοντέμ να εργαζόμαστε και έχουμε μεγάλες δυσκολίες και πρέπει λοιπόν όλα αυτά να αντιμετωπιστούν σε βάθος και άμεσα. Φυσικά έχουμε και τις αγορές online διαδικτυακά και εδώ πρέπει σε μεγάλο βαθμό στους πολίτες μας, στους καταναλωτές να δημιουργήσουμε ένα κλίμα εμπιστοσύνης ώστε να μπορούν να εμπιστεύονται και να αγοράζουν στο διαδίκτυο ηλεκτρονικά και υπάρχουν πολλές ανησυχίες και μελήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Αν δούμε κυρίως τι προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη στρατηγική της και τι έχει ενταχθεί σε αυτήν. Και θέλουμε να δούμε, πραγματικά θα έχουμε διαφορετικούς κανόνες και κανονισμούς ανάλογα με το αν αγοράζουμε offline ή online, διαδικτυακά ή εκτός διαδικτύου. Θα έχουμε διαφορετικούς κανόνες όταν θα αγοράζουμε ψηφιακά και εκτός ψηφιακών διαδικασιών. Ποιες διαδικασίες θα ισχύουν διασυνοριακά και εκτός διασυνοριακών αγορών. Η απάντηση είναι σαφής. Δεν μπορούμε τέτοιου είδους κατακαιρματισμένες ρυθμίσεις να έχουμε. Πρέπει να εξετάσουμε πολύ προσεκτικά τι προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτόν τον τομέα σφαιρικά. Και έχουμε και τον τομέα που είναι πολύ σημαντικό, το πρόβλημα του geo-blocking της ε, φραγής ε, ε, ή των γεωγραφικών ορίων φραγών και στον ψηφιακό τομέα, στο geo-blocking, δεν έχουμε κάνει πολλά πράγματα, διότι αυτά είναι θέματα της Επιτροπής Πολιτισμού. Αλλά το geo-blocking στις αγορές ε, online, διαδικτυακά, βλέπουμε ότι μπορεί κάποιος ή θέλει να αγοράσει σε μια ιστοσελίδα και αυτόματα τον μεταθέτουν σε μια άλλη, τον περνάνε αμέσως σε μια άλλη διότι υπάρχει άλλη ηλεκτρονική διεύθυνση σε άλλη χώρα. Αυτά είναι θέματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν και πρόκειται και για θέματα ανταγωνισμού που πρέπει να ρυθμιστούν επίσης στις πλατφόρμες. Πρέπει να σκεφτούμε να δούμε πώς θα μεριμνήσουμε τα ψαχτήρια, οι μηχανές έρευνας, έρευνας να διασφαλίζουν ισοδίκαιο ανταγωνισμό με τα ψαχτήρια. Πώς μπορούμε να το προωθήσουμε αυτό και στον τομέα της επιμεριζόμενης κοινή οικονομίας, sharing economy, να δούμε ποιες επιπτώσεις έχουν όλα αυτά. Θέλουμε επισφαλείς, πολλές επισφαλείς, μη ασφαλείς θέσεις εργασίας ή θέλουμε κανόνες και κανονισμούς. Η Καλιφόρνια είναι ένα καλό πρότυπο, ένα καλό παράδειγμα για μας. Και μια και βλέπουμε ότι ο χρόνος πιέζει πάρα πολύ βέβαια και περνάει, είναι ένα πολύ ευρύ θέμα αυτό, η οικονομία δεδομένων, η ουδετερότητα μεροληψία του δικτύου, η ηλεκτρονική διαχείριση και διακυβέρνηση, e-governance και για το αν είμαστε όλοι μια άποψη ή όχι, συνενετικά ή όχι, όλα αυτά πρέπει να τα συζητήσουμε και πολλά θα είχα να πω ακόμα. Ευχαριστώ. Uh, thank you very much, Ευχαριστούμε πολύ. Ευτυχώ έχετε και την ε, συνεισηγήτρια. Επομένω μπορεί εκείνη να προσθέσει όσα εσείς ε, παραλείψατε. Κυρία Κάλλα, ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και εγώ για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε με την κυρία Γκέπχαρτ και για αυτό το φάκελο. Ανέφερε και η ίδια ότι δεν ήταν ε, εύκολος ο φάκελος αυτός. Σε κάποια ζητήματα διαφωνήσαμε, όμως τελικά λειτουργήσαμε και εξισορροπητικά, αν θέλετε. Γενικά είναι πολύ σημαντικό οι δύο κοινοβουλευτικέ επιτροπέ να εξακολουθήσουν να συνεργάζονται και να οικοδομούν την αμοιβή αυτή εμπιστοσύνη. Γιατί βλέπουμε ότι σε πολλά θέματα είναι αρμόδιες και πολλές άλλες επιτροπές και πρέπει να τα λάβουμε όλα αυτά υπόψη. Για το χρονοδιάγραμμα αρχικά λάβαμε έτοιμα και από το ΕΛΚ να μετατεθεί ψηφοφορία από τις 11 στις 14 μπορώ να δεχθώ αυτό το αίτημα, αν υπάρχει πολιτική στήριξη και από όλε τι πολιτικέ ομάδε, η έκθεση να πάει στην Ολομέλεια τον Ιανουάριο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί όλοι έχουμε συμφωνήσει επί ενό χρονοδιαγράμματο ε, για να εκπονηθεί μια έκθεση γρήγορα, ώστε και το θεσμικό μα όργανο να έχει λόγο στην όλη διαδικασία όταν ξεκινήσει η νομοθετική πρωτοβουλία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ψηφιακή ενιαία αγορά. Για την ίδια την έκθεση θα επικεντρωθώ στα πιο σημαντικά ζητήματα από πλευρά ΙΤΡΕ. Ε, Ήθελα να μεταφέρω το βασικό μήνυμα ότι αν η Ευρώπη αποτύχει και δεν καταφέρει μάλλον να στρέψει προς το όφελός της αυτή την ψηφιακή επανάσταση, τότε οι απώλειες μπορεί να είναι τεράστιες αυτές οι καινοτομίες και οι νέες τεχνολογίες είναι πραγματικά κέρια σημασίας για την ανταγωνιστικότητα και τις οικονομίες μας. Πάντα αναφέρομαι, ε, για παράδειγμα, στον ε, αργαλιό, όπως παλιότερα υπήρχε αυτή η διαμάχη για το αν θα χρησιμοποιείται ή όχι. Δεν έχει νόημα να κάνει κάποιος αυτή τη διαμάχη όταν έχει ήδη εφευρεθεί η ε, συσκευή, η μηχανή. Πρέπει λοιπόν να περάσουμε στην αξιοποίηση αυτών των μέσων. Η νέα ψηφιακή αγορά θα πρέπει να διαμορφώσει νέα κλίμακα για τις ε, επιχειρήσεις στην Ευρώπη. Από τις πολύ μικρές μέχρι τις μεγαλύτερες. Γι' αυτό θέλουμε και ένα πλαίσιο και μια πολιτική ε, φιλική προς ε, την καινοτομία για τις πλατφόρμες που να δημιουργεί νέες ευκαιρίες. Να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα για τις επιχειρήσεις. Ο χρήστη βεβαίω είναι πολύ σημαντικό στοιχείο τη όλη διαδικασία, κινητήριο δύναμη. Γι' αυτό και θέλουμε μια στρατηγική με ενεργού ε, πολίτε και καταναλωτέ ε, και δυνατότητα μεταφορά των δεδομένων, αλλά και ιδιοκτησία των δεδομένων. Η ανάπτυξη δεν προκύπτει μόνο από τον τομέα ε, της τίμης τεχνολογίας, αλλά και από τις επιμέρους, από την αξιοποίηση των τεχνολογιών ACT από άλλες βιομηχανίες και η βιομηχανία δηλαδή εν γέννη μπορεί ε, να υποφεληθεί από την ε, υιοθέτηση ψηφιακών τεχνολογιών. Και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να κάνει μία αναθεώρηση για τα μεγάλα δεδομένα, τα big data, ε, πώς θα διαμορφωθεί μία ψηφιακή αγορά για το διαδίκτυο που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή και να έχει ως στόχο αυτή την πρωτοβουλία για την ελεύθερη ροή δεδομένων και την άρση φραγμών και περιορισμών. Επειδή δεν υπάρχει αυτή η ενιαία αγορά για τα δεδομένα, δεν έχει πλέον νόημα για τις επιχειρήσεις να επενδύουν σε αυτές τις μεγάλες κλίμακας ε, προγράμματα. Και κάποια άλλα στοιχεία είναι πολύ σημαντικά για την καινοτομία. Πρώτον, οι υποδομές η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλει να διασφαλίσει ότι διατηρείται η ανταγωνιστικότητα και διαφυλάσσει την ανταγωνιστικότητα στην αγορά τηλεπικοινωνιών με πρόσβαση στην αγορά και με ομοιόμορφη εφαρμογή των κανόνων. Η ενιαία ρυθμιστική αρχή τηλεπικοινωνιών δεν αντικαθιστά τι εθνικέ αρχέ. Βεβαίω και θα πρέπει να παραμείνουν εθνικέ αρχέ. Όμω η ενιαία αυτή ρυθμιστική αρχή θα μπορούσε να έχει μια πληρέστερη εικόνα ε, ολόκληρου του κλάδου των τηλεπικοινωνιών. και έτσι θα μεριμνά του ώστε κανεί να μην προσπαθεί να προστατεύσει μόνο τη δική του αγορά. Και θα έχει και την κατάλληλη εποπτεία της ενιαίας αγοράς. Αυτό συνδέεται και με την διασφάλιση της αρχής ε, της ουδετερότητας του διαδικτύου και της ε, ομοιόμορφης εφαρμογής αυτής της αρχής σε όλη την Ευρώπη αλλά συνδέεται και με την ε, κατάργηση των ε, τελών περιαγωγής. Και τέλος, έχουμε και τον ρόλο της δημόσιας διοίκησης και των κυβερνήσεων, που είναι εξαιρετικά σημαντικός σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί αυτό ξεκινάει από, τα, την ε, δημοσίευση ανοιχτών δεδομένων μέχρι και με την ε, καινοτομία είναι σημαντικό για τις μικρές επιχειρήσεις για να βρουν νέες λύσεις. Αλλά και η ηλεκτρονική διακυβέρνηση και άλλα μέσα ε, για να διευκολύνουμε τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να εξοικονομήσουμε χρόνο και αυτό γενικά θα μας διευκολύνει να ασχοληθούμε με ό,τι ασχολείται ο καθένας. Το ανέφερε η κυρία Γκέπχαρτ ότι δεν συμφωνούμε με αυτή την ε, αρχή άπαξ, όμως ε, εγώ τη στηρίζω στην αρχή, γιατί οι επιχειρήσεις μπορούν ε, πραγματικά να κερδίσουν πολύ χρόνο αν δώσουν τα δεδομένα μόνο μία φορά και τέλος. δεν χρειάζεται να υπάρχει και πολλή γραφειοκρατία. Αυτά είναι τα κύρια ζητήματα που θέλω να θίξω, αν και υπάρχουν και άλλα ε, που εντάσσονται σε αυτή την έκθεση. Όμως περιμένω να ακούσω και τα δικά σας σχόλια, τις γνώμες σας, αλλά και προσβλέπω σε αγαστή συνεργασία με τους συναδέλφου. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Και οι δύο συνεισηγητρίες θα έχετε δυνατότητα να πάρετε το λόγο και στο τέλος για κάποια καταληκτικά σχόλια. Αρχικά θα ήθελα να πω ότι η πρόταση για τις 14 Δεκεμβρίου να γίνει τότε ψηφοφορία είναι Δευτέρα βράδυ στο Στρασβούργο. Είναι νομίζω μια καλή πρόταση. Αλλά πρέπει να υπάρχει στήριξη από όλες τις πολιτικές ομάδες. να συμφωνήσουν ότι θα ψηφίσουμε τον Ιανουάριο. Η σύσταση από τη ε, διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών. Μπορούμε να προσπαθήσουμε με την κυρία Βίκη Φόρτερ να στηρίξουμε αυτή την πρόταση και να πάμε στη διάσκεψη των Προέδρων. Επομένω, προ του ε, συντονιστέ και των δύο επιτροπών να Παρακαλώ να έχετε κατά νου αυτό το στοιχείο. Ότι αυτές οι δύο ημερομηνίε, Ιανουάριο στην Ολομέλεια και πιο πριν, 14 Δεκεμβρίου, Δευτέρα στο Στρασβούργο, ψηφοφορία και στις δύο επιτροπές. Και τώρα περνάμε στους ε, σκιώδεις ή στους αναπληρωτές. Τρία λεπτά έκαστος. Θα αναβήρκουνεν από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τις δύο εισηγήτριες. Ευχαριστώ, κυρία Κάλλας και κυρία Κεπχάρτ. Είναι πολύ σημαντική αυτή η έκθεση. Ξέρουμε ότι μια ευμερούσα ενιαία ψηφιακή αγορά στην Ευρώπη είναι πραγματικά κραγωνιά λήθο ε, για την οικονομία και, την απασχόληση στην Ευρώπη, αλλά και για τον εξυγχρονισμό τη παραδοσιακή βιομηχανία. Δεν έχουμε ακόμα όμω την ενιαία ψηφιακή αγορά. Οι φραγμοί μεταξύ 100 μελών θα πρέπει να αρθούν για να υπάρξει μια πραγματικά ενιαία ψηφιακή αγορά. Θέλουμε να προσφέρουμε στους πολίτες μας μια μεγαλύτερη ποικιλία ε, δεσυνοριακών ε, υπηρεσιών με ανταγωνιστικές τιμές και να διευκολύνουμε την πρόσβαση στις επιχειρήσεις και ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε ό,τι αφορά τις δεσυνοριακές αγορές. Ξέρουμε ότι οι νέε υπηρεσίε μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο όταν υπάρχει ευρύτατη και αξιόπιστη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Γι' αυτό πρέπει να διασφαλίσουμε και να ενισχύσουμε τις επενδύσεις στι υποδομές, ιδίω ό,τι αφορά τα νευροζωνικά δίκτυα. Όλοι οι πολίτες θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ψηφιακή οικονομία, δική μας ε, ευρωπαϊκή βιομηχανία θα πρέπει να είναι παγκοσμίω ανταγωνιστική. Θέλουμε να έχουμε αποφάσεις πλαίσιο που να ενθαρρύνουν και να διευκολύνουν ε, τις ε, επιχειρήσεις τηλεπικοινωνιών να γίνουν πανευρωπαϊκέ. Σας ευχαριστώ λοιπόν για αυτό το προσχέδιο έκθεσης. Νομίζω ότι αποτελεί μια καλή βάση για τις μελλοντικέ ε, εργασίε των εισηγητριών και των σκιωδών να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Κάτι το οποίο θα θέλαμε εμείς να ενισχύσουμε μέσα στην έκθεση είναι η βιομηχανική βάση της. Και αυτό είναι λογικό γιατί προερχόμαστε από την Επιτροπή ακριβώ Βιομηχανία, Έρευνα και Ενέργεια. Υπάρχουν δύο σκέλη όταν εξετάζουμε την ψηφιοποίηση και τη βιομηχανία. Αφενό, πρέπει να εξετάσουμε πώς θα επιταχύνουμε την ψηφιοποίηση της ίδια βιομηχανίας. Και αυτό αφορά και την παραδοσιακή βιομηχανία, αλλά και άλλε πλευρές βιομηχανίας... Όπω είναι κατασκευέ, ενέργεια, μεταφορέ, ελληνικό εμπόριο, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες ε, και εκπαίδευση. Όλα αυτά πρέπει να ενισχυθούν. Και δεύτερον, πρέπει να δούμε πόσο η βιομηχανία μπορεί να βοηθήσει ε, και να ενδυναμώσει την διαδικασία ψηφοποίηση στην κοινωνία. Γιατί έτσι έχουμε και νέα επιχειρηματικά μοντέλα και νέε υπηρεσίε. Όλα αυτά βοηθούν την ε, αύξηση τη απασχόληση και τη δημιουργία θέσεων εργασία. Ξέρουμε ότι πολλέ ε, μεταρρυθμίσει θα πρέπει να γίνουν για την ανάπτυξη τη ενιαία ψηφιακή αγορά και ε, για να μπει η Ευρώπη στην ψηφιακή εποχή. Σε πολλέ περιπτώσει πρέπει να αλλάξουμε την οτροπία ότι ο ψηφιακό κόσμο θα είναι διαφορετικό ε, ή θα είναι ξεχωριστό από τον κανονικό κόσμο. Αντιθέτω, πρέπει να διασφαλίσουμε ένα ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού και για τις ψηφιακές και για τις παραδοσιακές ε, δομές. Θεωρούμε ότι υπάρχουν πολλές ευκαιρίες από την ψηφιοποίηση και θέλουμε να υπάρξει περαιτέρω συνεργασία με όλους σας. Σας ευχαριστώ και άλλος εκπρόσωπος τώρα από το ΕΛΚ, Φιλίπ Σουδά. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, καταρχάς να συγχαρώ με τη σειρά μου τις δύο συνεισηγήτριες Γκέμπερτ και Κάλλας για τα ευθύ κείμενα που συνέταξαν θα είναι πολύ πιο εύκολο να τροποποιηθούν διότι ακριβώς είναι ευθύ. Η Ευρώπη έχει καθυστέρηση διότι ξέρουμε ότι μεγάλο ποσοστό της τεχνολογίας προέρχεται από τις ΗΠΑ και αν θέλουμε να ε, ε, γίνουμε μια δύναμη θα πρέπει να αναπτύξουμε περαιτέρω το, το μοντέλο μας. Θα πρέπει να ε, επηρεάσουμε και να μετατρέψουμε όλη την οικονομία μας σε ψηφιακή οικονομία. Δεν πρόκειται μόνο για την βελτίωση των νέων τεχνολογιών, αλλά την μετατροπή όλη της παραδοσιακής οικονομίας σε ψηφιακή οικονομία. Πρέπει να ευνοήσουμε τα νέα οικονομικά μοντέλα όπως αυτό του επιμερισμού σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο και να μπορέσουμε να μετατρέψουμε τη γνώση σε χρυσό. Κάνουμε λοιπόν την Ευρώπη μια, μια ισχύ ψηφιακή, διότι μόνο έτσι θα μπορέσουμε να επικρατήσουμε. Διαφορετικά οι υπόλοιποι θα μας ξεπεράσουν και η κατάστασή μας θα είναι πολύ πιο δύσκολη. Και δεν πρόκειται να τους ε, φτάσουμε. Πρώτα απ' όλα νομίζω ότι τα νομικά καθεστώτα θα πρέπει να προσεγγίσουν τα μεν τα δε ανάμεσα στην ε, επιγραμμική πώληση και μη επιγραμμική πώληση. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να προσαρμόσουμε. Δεύτερον, χρειάζεται η κίνδυνη σε ό,τι φορά την ευθύνη αλλά και ε, τον επιμερισμό των ε, τόσο δαπανών αλλά και των κερδών θα πρέπει να είναι απόλυτα σωστά επιμερισμένα θα πρέπει να καταλήξουμε σε ένα σύστημα το οποίο θα είναι αξιόπαστο, νόμιμο, δίκαιο και έχω υπόψη μερικές πλατφόρμες. Τρίτον, θα πρέπει να ε, ανακαλύψουμε ένα νέο φορολογικό σύστημα. Με λίγα λόγια θα πρέπει να ε, ε, εφευρέσουμε την ΦΠΑ του 21ου αιώνα, δηλαδή δεν υπάρχει ΦΠΑ που θα εφαρμόζεται σε μια παρόμοια οικονομία. Τέταρτον, ε, η γνώση και η δημιουργία, η ευρηματικότητα θα είναι σημαντικέ. Θα πρέπει να στηρίξουμε λοιπόν αυτή την ευρηματικότητα, αυτή τη δημιουργικότητα και πέμπτον, θα πρέπει να ασφαλίσουμε ότι οι υποδομέ θα αναπτυχθούν, θα εξελιχθούν. Δεν μπορεί να υπάρξει ψηφιακή οικονομία δίχω κατάλληλη υποδομή. Και παντού ο κανόνα θα πρέπει να είναι απόλυτο, θα πρέπει να σιωπήσουν τα εθνικά συμφέροντα και να έχουμε ένα οικονομικό σύστημα που είναι πραγματικά ευρωπαϊκό, ενωσιακό και όχι καραγερματισμένο ανάμεσα σε 28 κράτη. Αυτά, Πρόεδρε, πολύ μίλησα. Η Ευρώπη σε πολλές βιομηχανικές επαναστάσεις. Ε, ανακαλύψαμε την τυπογραφία, τον, ε, την, ε, αερο, αεροπορική βιομηχανία, την αυπηγική. Σε όλες αυτές τις εξελίξεις η Ευρώπη δεν ήταν η, αυτή που εφήβρε τα πάντα. Θα πρέπει λοιπόν διαδραματίσουμε έναν σημαντικό ρόλο, διαφορετικά θα, μας, θα μείνουμε στην γωνία. Ευχαριστώ συνάδελφοι, κυρία Νάτσολη από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Ευχαριστώ, χαίρομαι που δουλεύω επί του ζητήματος αυτού και θα είναι πολύ καλή ιδέα 120 από εμά να δουλέψουμε πάνω σε αυτό. Ε, λάβαμε διάφορες απόψεις από επιτροπές και θα πρέπει σε αυτού του να ανταποκριθούμε στις, ε, σε αυτά τα οποία μας ζήτησε η Κομισιόν ειδικά με την ψηφιακή οικονομία, κοινωνία, συγγνώμη. Είναι σημαντικό να προχωρήσουμε τις επενδύσεις, διότι δεν υπάρχει ψηφιακό μέλλον για την Ευρώπη αν υπάρχει ένα ψηφιακό χάσμα. και κάποιες μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μην είναι σε θέση να ακολουθήσουν τις εξελίξεις. Θα πρέπει να πούμε στους εμπλεκόμενους τι θα πρέπει να πράξουν, αλλά και όχι μόνο. Όταν λοιπόν Υπάρχουν κάποιες αποτυχίες θα πρέπει να προχωρήσουμε, να βοηθήσουμε κάποιες περιφέρειες. Ο δεύτερος πυλώνας ε, για την ψηφιοποίηση είναι, είναι η εμπιστοσύνη στις υπηρεσίες αλλά και στις τονολογίες. Κάθε φορά προκύπτουν νέες λύσεις, η ασφάλεια είναι κάτι το πολύ σημαντικό και όσο περισσότερο Προγράμμι στην ψηφιοποίηση, τόσο μεγάλη προσοχή πρέπει να δίνουμε σε αυτά τα ζητήματα. Τώρα το ζήτημα της ασφάλειας, ε, της ε, ιδιοκτησίας των ε, στοιχείων, δεδομένων κλπ. Χθε είχαμε συζητήσεις στην Επιτροπή μας και τα συμπεράσματα ήταν αρκετά ενδιαφέροντα. Δεν πρόκειται για εξέλιξη και επανάσταση της ονολογίας, αλλά είναι το κοινωνιακό πρότυπο που επιλέγουμε μετά από την ψηφιοποίηση. Εργαζόμαστε λοιπόν και πάνω σε αυτό το ζήτημα, αλλά θεωρώ ότι θα πρέπει να γνωρίζουμε πώς θα επηρεαστεί το κοινωνικό μοντέλο και τι κοινωνικό μοντέλο θέλουμε να δημιουργήσουμε. Οι αλλαγές θα γίνουν, αλλά εμείς είμαστε υπεύθυνοι για την ε, συγκρότηση της κοινωνίας και δεν θα πρέπει να μας φοβίζουν οι πλατφόρμες. Υπάρχουν πολλά είδη, υπάρχει βιομηχανική πλατφόρμα, υπάρχουν ζωτική σημασία πλατφόρμας και η ακρόαση της Επιτροπής είναι πολύ ενδιαφέρουσα, αλλά είναι δύσκολο εάν ακούνε μόνο τις τηλεπικοινωνίες Καταλήγω λοιπόν ε, το θέμα του διεθνούς ανταγωνισμού, το 5G. Πρέπει λοιπόν να είμαστε να γίνουμε πρώτοι και όχι ουραγοί της όλης διαδικασίας. Ευχαριστώ. Δύο εκπρόσωποι τώρα της ECR ε, έχουν το λόγο, η κυρία Βεκή. Ευχαριστώ. Είμαι από την του. Γιατί τα κάνουμε όλα αυτά, διότι η ψηφιακή αγορά είναι μια αγορά πολύ σημαντική και μπορεί να βοηθήσει στην ε, αναπασχόληση και την ανάπτυξη. Και αυτό είναι ο πυρήνας των ζητημάτων που εξετάζουμε στην Επιτροπή μας δύο κρατήδες αρχές. Πρώτα απ' όλα ότι το ζήτημα αυτό έχει, παρουσιάζει ιδιαίτερη υψηλή ταχύτητα. Οι εξελίξεις είναι ταχύτατες. Κοιτάζουμε το μέλλον και δεν θα πρέπει να παραμείνουμε μόνο στο πλαίσιο μονοπόλιο. Δεύτερον, οι ψηφιακές αγορές δεν έχουν όρια, δεν έχουν περιθώρια. δεν γνωρίζουν σύνδερα με λίγα λόγια. Έχω, κατα... έχω καταρτήσει πολλές τροπολογίες μαζί με άλλους συναδέλφους άλλων επιτροπών και θέλουμε να ε, εξετάσουμε το ζήτημα σφαιρικά. Καταρχήν για το ηλεκτρονικό εμπόριο υπάρχουν τομείς για την οικοδόμηση εμπιστοσύνη των κανολτών στο ε, ηλεκτρονικό εμπόριο όπως την κατάργηση πολλών ε, διαδικασιών που χρειάζονται ε, έντυπα νομίζω πως υπάρχουν και ζητήματα τα οποία έχουν με, να κάνουν με την ασφάλεια των πληρωμών στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου και αυτά τα θέματα πρέπει να μας απασχολήσουν τα δικαιώματα των καταναλωτών. Υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στα ψηφιακά αγαθά και τα, τα ε, υλικά αγαθά. Όταν λοιπόν κοιτάζουμε, εξετάζουμε αυτά τα ζητήματα θα πρέπει να εντοπίσουμε τις διαφορές που υπάρχουν και πού μπορεί να πετύχουμε τις κατάλληλες ε, αλλαγές στις νομοθεσίες τώρα για τα προδοσιακό εμπόριο, ε, αγορές, συγγνώμη. Όταν ε, θα πρέπει να, εξετάσουμε, πρέπει να τα εξετάσουμε παράλληλα. Υπάρχουν χώρες όπου ε, η Κομισιόν έχει ζητήσει να αναλυφθούν κάποιες δράσεις ε, αναφορικά με τις βέλτιστες πρακτικές. Θα πρέπει να δούμε τι θα πρέπει να γίνει μετά από τις νομοθεσίες top-down για το geo-blocking χρειάζεται να επιλύσουμε τα πραγματικά προβλήματα για τους καταναλωτές έχω καταναλώσει ο χρόνο ομιλίας μου θα, θα είμαι σύντομη ε, διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν διαφορετικέ τιμέ και εδώ ε, έχει, υπάρχει και το άρθρο 20 της, οδη, της οδηγίας περί ε, καταναλωτών, περί πεσίων, συγγνώμη. Και υπάρχει και το ζήτημα του ανταγωνισμού και θα πρέπει να ε, διασφαλίσουμε ότι έχουμε καλύτερη πρόσβαση και όταν θέτουμε κάποια πρότυπα να μην δημιουργούμε παράλληλα ε, νέα μονοπόλια. Ευχαριστώ. Καταλαβαίνω ότι, καταλαβαίνετε ότι ήταν πολύ δύσκολη η θέση μου, παρατηρεί ο Πρόεδρος, αλλά νομίζω πως θα επιζήσουμε όλοι μας. Τώρα πλευράς ECR, ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Hans Βόλαφ. Θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα σημείο μόνο, το οποίο είχε προαναφερθεί, όμως που πολύ στεναρά πιστεύω ότι είναι σημαντικό. Φυσικά πρέπει να υποβάλουμε προτάσεις και συστάσεις, όμως θα πρέπει επίσης να πούμε και τι δεν πρέπει να πράξουμε. Και η εντύπωση που έχω αποκομίσει για αυτά τα οποία προετοιμάζονται τώρα σε αυτή τη φάση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι η εντύπωση ότι διανέμουμε, διαχέουμε στόχους που δεν είναι όλοι αναγκαίοι. Δεν τους χρειαζόμαστε. Πρέπει να επικεντρωθούμε στα θέματα που πολλά από αυτά έχουν ήδη παρουσιαστεί, που είναι ουσιώδη. Όμως, <clears throat> αναφέρει στόχους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το βαθμό, το ποσοστό των αγορών διαδικτυακά, ηλεκτρονικά. Για παράδειγμα, στην γερμανική αγορά ή στις γερμανικές επιχειρήσεις, οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Είναι περιττό, είναι άχρηστο να αποφασίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι μια χώρα θα ή στο 2020-2025 πάνω από το ίμιση των αγορών στο διαδίκτυο, διαδικτυακά, ηλεκτρονικά. Αυτό πρέπει να είναι η δουλειά των κρατών, των κρατών και δεν πρέπει να είναι αρμοδιότητα των θεμάτων που πρέπει να ρυθμίσουμε εμείς και η Επιτροπή. Λοιπόν, ζητώ να απορρίψουμε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσα στο πλαίσιο αυτής της έκθεσης. Thank ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, συνολικά βρισκόμαστε στα πλαίσια του χρόνου που έχουμε. Και τώρα ένας εκπρόσωπος της Άλντες και εισηγητή. εισηγητής. Χαράντσοβα. Δίτα Χαράντσοβα από την ΙΜΚΟ, παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα να ξεκινήσω ευχαριστώντας από πλευράς εισηγητών για αυτή την έκθεση. Ε, είναι μια πολύ ισορροπημένη έκθεση. Να τονίσω σύντομα τρεις κύριες αρχές που πρέπει να λάβουμε υπόψη όταν συζητάμε την ενιαία αγορά. Ρόλος μας πρέπει πρώτα να είναι να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο για αυτή την αγορά να μην ρυθμίσουμε κανονιστικά κάθε λεπτομέρεια και κάθε μικρό τμήμα. Δουλειά μας είναι να δημιουργήσουμε την μεγάλη ευρύτερη δομή στην οποία θα λειτουργήσει αυτή η αγορά. Αλλά να αφήσουμε ελεύθερους τους όσους θα εμπλακούν μέσα σε αυτό το ελαστικό ευλίγιστο νομικό πλαίσιο να δράσουν. Οι επιχειρήσεις θα αποφασίσουν πώς θα εφαρμόζουν αυτούς τους κοινού κανόνες και τις αρχές επί των οποίων θα έχουμε συμφωνήσει. Όταν θα έχει δημιουργηθεί όμω αυτό το πλαίσιο, εμεί ω νομοθέτες Πρέπει να αποστασιοποιηθούμε, να τους αφήσουμε τους εμπλεκόμενους να καθορίσουν το τι θα κάνουν. Δεν πρέπει να υποστηρίξουμε προτάσεις να υπάρξει υπερβολική ρύθμιση από τον έξω κόσμο στον ψηφιακό κόσμο. Το περίπλοκο περιβάλλον για τις ψηφιακές δράσεις αυτό θα σήμαινε ότι θα θέλαμε ε, να, θα πρέπει να αφήσουμε ελεύθερη την ευρωπαϊκή οικονομία στον ψηφιακό τομέα για να είναι δημιουργική. Δεύτερο, δημιουργώντας αυτό το πλαίσιο, το έργο μας πρέπει να υποστηρίζει την καινοτομία. Πρέπει να υποστηρίξουμε εκείνους τους Ευρωπαίους που δημιουργούν νέες πλατφόρμες στην ε, κοινή επιμεριζόμενη οικονομία γύρω μας Πρέπει να τους ε, συνδράμουμε, να τους υποστηρίξουμε καθώς δοκιμάζουν νέες ε, ιδέες οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί και οι οργανώσεις όπου δημιουργείται ένα νέο πολιτιστικό περιβάλλον χωρίς να κυλιδώνεται από, ε, ας το πω έτσι, μια προκατάληψη ή προκατηλημένη άποψη περί αποτυχίας όλοι ήταν παρόντες στην επιτροπή μας, στην επίσκεψη του Silicon Valley στην Καλιφόρνια και είδαμε ότι η ελευθερία καινοτομία είναι αυτή η οποία οδήγησε στην ψηφιακή επανάσταση εκεί. Μετά από αυτή την αποστολή μας είμαι πισμένη απόλυτα ότι δεν χρειάζεται να αποφύγουμε εξωτερικό ανταγωνισμό ή να δημιουργήσουμε ε, πρωταθλητές ευρωπαϊκούς. Αν κάποιος γίγαντας στον ψηφιακό, στον ψηφιακό κόσμο καταρρεύσει, αυτό θα σημαίνει ότι δεν υποστηρίχθηκε και δεν δημιούργησε το, το προϊόν το οποίο προτιμούν και επιλέγουν οι πολίτες. Και τέλος, όταν θα έχουμε τη δημιουργία αυτού του πλαισίου, πρέπει να βρούμε τρόπους να αρθούν τα προσκόμματα και τα εμπόδια τα οποία δημιουργούνται για αυτόν τον ψηφιακό κόσμο το geo-blocking και κανόνες πνευματικής ε, ή διανοητικής ιδιοκτησίας ε, για τα προϊόντα και τα δημιουργήματα, αλλά επίσης η ψηφιακή επανάσταση να εφαρμοστεί και για τις αρχές ε, και η παραγωγή να προαχθεί στις επιχειρήσεις και η ιδιωτική ζωή όλων των πολιτών να απλουστευτεί και να διευκολυνθεί. Σας ευχαριστούμε κυρία. Δύο εκπρόσωποι της ΓΚΟΕ της Ενωτικής Αριστεράς. Η κυρία Κορνέλια Έρνς πρώτη παρακαλώ από την Ήτρε. Σας ευχαριστώ θερμά και τις δύο εισηγήτριες ευχαριστώ θερμά φυσικά θα έλεγα, είναι σαφές ότι πρόκειται εδώ για ένα σημαντικό εγχείρημα, ένα σημαντικό χαρτοφυλάκιο. Και θέλω σε ένα σημείο <clears throat> να, να πω ότι έχουν δίκιο οι προλαλήσασες και οι προλαλήσαντες. Μάλιστα, πρέπει να υπάρξουν κανόνες και κανονισμοί. Εκεί όμως όπου χρειάζονται. Και όχι να ρυθμίζουμε επί παντός του επιστητού τα πάντα. Και σημαντικό είναι για μας να υπάρχει ισορροπία μεταξύ ανταγωνισμού αφενός και διασφάλισης θεμελιωδών δικαιωμάτων αφετέρου. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για μας. Πολλά μπορεί να κάνει κανείς και όσον αφορά τα δικαιώματα των αγοραστών για αγορές στο διαδίκτυο ηλεκτρονικά, αλλά όμως εδώ δεν είναι το θέμα μόνο προσαρμογής δικαιωμάτων, αλλά ενδυνάμωσης, ενίσχυσης δικαιωμάτων και δημιουργία κανόνων και κανονισμών για να είναι σαφές το πλαίσιο στο οποίο θα γίνεται αυτό. Και διαφάνεια των κανόνων και όσον αφορά τα πνευματικά δικαιώματα, το copyright. Τι είναι αυτά τα οποία επιθυμούμε και τι είναι αυτά τα οποία δεν θέλουμε να γίνουν. Σημαντικά είναι επίσης ως στοιχεία η κατάργηση των ε, geo-blocking. Δεν είναι καινούριο αυτό και πολλοί συνάδελφοι ανέφεραν παρόμοιες απόψεις από πλευρά τους προηγούμενα. Πρέπει να υπάρξει σαφήνεια εδώ που θα δημιουργήσουμε και αυτό είναι ένα σημείο επί του οποίου θα δράσουμε εντονότερα. Τώρα, κάτι άλλο. Ε, ε για όλες εκείνες τις προσδοκίες και όλες τις ρυθμίσεις η αρχή της ουδετερότητας αμεροληψίας του δικτύου δεν πρέπει να θυγεί, δεν πρέπει να αλλοιωθεί. Πρέπει να υπάρχει ελευθερία προσπελασιμότητας πρόσβασης στα δεδομένα, στο διαδίκτυο, με ίσους όρους και προϋποθέσεις για όλους. Το θέμα της ουδετερότητας του δικτύου δεν μπορεί να είναι ένα θέμα το οποίο ε, θα εμπλέκεται όσον αφορά την κατάργηση των ε, τελών περιαγωγής. Και πρέπει να είμαστε συνεπείς σε όλα αυτά και είναι σημαντικό αυτό. Επίσης είναι σημαντικό όταν κάνουμε λόγο για την ανάπτυξη υποδομών που είναι πολύ σημαντική υπόθεση, αδιαμφισβήτητα πρέπει να υποστηριχθεί η ενδυνάμωση, η ενίσχυση των υποδομών και η ασφάλεια των δεδομένων. Είναι πολύ σημαντική υπόθεση. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε την ομολογία, την απόφαση του ΔΕΚ, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, για το Safe Harbor και αυτό θέτει εδώ τους φραγμούς και τα όρια. Δεν μπορούμε να παρακάμψουμε αυτή την αρχή υπάρχει δικαίωμα για την αυτοδιάθεση των δεδομένων των πολιτών. Και εδώ δεν υπάρχουν ε, δυνατότητες να υπονομευθεί, να παρακαμφθεί αυτή η αρχή. Και αντίστοιχα με τροπολογίες θα καλύψουμε αυτό το πεδίο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος. Και εξ ονόματος ε, πάλι της Γκουεπα τώρα. Ντένις Ντε από την ΙΜΚΟ παρακαλώ. Ο κύριος Ντε Δεν uh, παρίσταται. Προχωράμε. Πάμε παρακάτω. Δύο εκπρόσωποι τώρα των Πρασίνων του πολιτικού, uh, της πολιτικής ομάδας των Πρασίνων. Από την Ήτρε, εσείς παρακαλώ, δεν ο εκπρόσωπος των Πρασίνων. Η κυρία από πλευρά σας τη ΣΥΜΚΟ Ρέντα παρακαλώ. take, uh, minutes, but... Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη και να μην καλύψω όλο το χρόνο. Πρώτον, η, η συγγήτρια και συνεισηγήτρια, η κυρία Γκέπαρτ και Κάλλας, έκαναν εξαιρετική δουλειά μέχρι σήμερα. Το σχέδιο δίνει μια σημαντική γραμμή αφετηρίας για τις διαβουλεύσεις μας και συμφωνούμε απόλυτα με την γενική κατεύθυνση της ε, ε, εργασίας αυτής. Οι ηλεκτρονικές ε, δραστηριότητες πρέπει να ενθαρρύνουν τον ανταγωνισμό και να ενδυναμώνουν τα θεμελιώδη δικαιώματα. Θέλω κάποιους τομείς να αναφέρω που πιστεύω ότι πιο λεπτομερώς, πιο εξειδικευμένα πρέπει να έχουμε κάποιες προσθήκες και όχι τόσο κάποιες ριζικές μεταβολές αυτού του σχεδίου. Πρώτον το ρυθμιστικό πλαίσιο των πλατφορμών ενώ συμφωνούμε με αυτά τα οποία έχουν γραφεί για το θέμα, πρέπει να αποστασιοποιηθούμε λίγο και να δούμε τα θεμελιώδη αυτά θέματα. Μέχρι σήμερα κανείς δεν μπόρεσε να μας επεξηγήσει τι είναι ουσιαστικά μια τέτοια πλατφόρμα. Και δυστυχώς ο ορισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως δόθηκε στις διαβουλεύσεις, δεν αποσαφηνίζει τα πράγματα. Είναι ένα μείγμα υπηρεσιών στο διαδίκτυο ηλεκτρονικά και μείγμα υπηρεσιών παρόχων. Και όλα τα παραδείγματα που δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι παραδείγματα ε, επιχειρήσεων όμως ε, δεν υπάρχει εδώ πιο εξειδικευμένη ρύθμιση. Ο ορισμός θα μπορούσε να σημαίνει ότι η δική μου ιστοσελίδα που έχει και κάποια διαφήμιση επάνω της μπορεί να θεωρείται και όλας πλατφόρμα. Ε, δεν γίνεται αυτό. Να, να επανεξετάσουμε όλα αυτά και να δούμε αν αυτή η ισοπεδωτική προσέγγιση one size fits all, δηλαδή ένα μέτρο θα καλύπτει τα πάντα, αν αυτό είναι το πιο ενδεδειγμένο και είδα προβλήματα σε σχέση με μια επιχείρηση που αναλαμβάνει ευθύνες σήμερα όσον αφορά το κοινωνικό δίκτυο Twitter και καταργούνται λογαριασμοί χρηστών όπου υπάρχουν κάποια κινούμενα σχέδια όσον αφορά και ε, ποδοσφαιρικά παιχνίδια. Όμως όλοι το κάνουν αυτό και όποιος έχει ένα λογαριασμό σε κοινωνικά δίκτυα, ο οποίος καταργείται και τον χρησιμοποιεί αυτόν και στην επαγγελματική του δουλειά, ε, είναι πολύ σοβαρή αυτή η ποινή, αυτό το πλήγμα. Πρέπει να είμαστε σαφείς, να σεβόμαστε τα δικαιώματα αυτών που χρησιμοποιούν αυτά τα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης, τα κοινωνικά δίκτυα. Ήδη έγιναν παρατηρήσεις για την αγορά ψηφιακού περιεχομένου και βλέπουμε ότι έχουμε και προσδοκίες χρηστών όταν ένα ηλεκτρονικό βιβλίο όταν αγοράζεται θεωρείται υπηρεσία ενώ ένα βιβλίο ως βιβλίο θεωρείται αγαθό. Πρέπει να δούμε τις διαχωριστικές γραμμές και να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε ένα πλαίσιο όπου ηλεκτρονικά, ψηφιακά θα μπορούν ως προϊόντα να αντιμετωπίζονται αυτά τα ε, αγαθά και όχι ως υπηρεσίες απλώς ε, διαδικτυακά. Πρόεδρος Διακόπτη, ευχαριστώ κυρία μου. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Ρέμον που αντι, ε, αν, αντικαθιστά τον κύριο Φάραντς, παρακαλώ. Um, Όπως είπαμε, υπό το πρίσμα των πρασίνων, η έκθεση αυτή όσον αφορά την ΙΤΡΕΠ ε, βαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση. Διαρωτώ πόσο σοβαρά παίρνουμε τον εαυτό μας και το έργο μας με τα ωραία λόγια που βρίσκουμε ότι ε, εδώ έχουν συγγραφεί. Στο σημείο 22 αναφέρεται ότι η ουδετερότητα του δικτύου είναι ένα σημαντικό στοιχείο στην ενιαία εσωτερική ψηφιακή αγορά και σε λίγες εβδομάδες θα ψηφιστεί προς έγκριση και για την κατάργηση της ε, ουδετερότητας στο διαδίκτυο. Αν εμείς πούμε ότι είναι σημαντική η ουδετερότητα του δικτύου αλλά την καταργήσουμε πιο πριν ψηφίζοντας κατά, ε τότε δεν είμαστε αξιόπιστοι. Στη συνέχεια, όταν έχουμε κάποιους παρόχους που μπορούν δωρεάν ε, κάποια περιεχόμενα στις τηλεπικοινωνίες να τις παρέχουν και όταν έχουμε ξεχωριστά τιμολόγια και αυτοί οι πάροχοι μπορούν δωρεάν να χρησιμοποιούν κάποια προϊόντα, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι όλοι οι μεγάλοι πάροχοι και ιδίω είναι Αμερικανοί πάροχοι αυτή τη στιγμή στο διαδίκτυο, θα έχουν πολύ μεγάλα προτερήματα και οι μικρές ευρωπαϊκές startups εταιρείες δεν θα μπορούν να ανταγωνιστούν. Αν τέτοια πράγματα αποφασίσουμε εμείς ως Ήτρε και στην Ολομέλεια είναι μόνο κενά ωραία λόγια και θα καταργήσουμε όλα όσα θέλουμε να πετύχουμε. Και για το geo-blocking και άλλες ε, τέτοιες προτάσεις που θέλουμε να υπερασπιστούμε και θεωρούμε ότι είναι σημαντικές, αν καταργηθούν όλη αυτή η έκθεση χάνει το περιεχόμενό της. Βρίσκω ότι η έκθεση αυτή είναι καλή και προχωρεί προς την σωστή κατεύθυνση. Να πάρουμε όσο στα σοβαρά τον εαυτό μας και τα λόγια μας και να είμαστε συνεπείς στις δράσεις μας, στα όσα εγκρίνουμε και ψηφίζουμε υπό αυτό το πνεύμα έτσι πρέπει να δράσουμε. Διαφορετικά θα είναι κενά περιεχομένου ωραία λόγια. Ευχαριστώ. E uh, Σας ευχαριστώ. David Μπορέλη από την Ήτρε, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τις εισηγήτριες Κάλλας και Γκέμπαρτ για την εργασία τους και για την πληρότητα της έκθεσης, η οποία είναι ιδιαίτερα ρεαλιστική. Θα επιθυμούμε να συμβάλλουμε για να διευρυνθεί η προσέγγιση με ένα βλέμμα το οποίο θα ατενίζει στο μέλλον. Βασικά είναι τρία τα σημεία ε, στα οποία θα επικεντρώσω την προσοχή μου. Είμαστε πεπισμένοι ότι κατά την υλοποίηση της ενιαία ψηφιακή αγοράς οι πολίτες θα πρέπει να τεθούν στο επίκεντρο. Δηλαδή η ψηφιακή, η ψηφιακή υπηκότητα θα πρέπει να ε, οδηγήσει σε μια ενεργό συμμετοχή των πολιτών στην ε, επιμερισμένη οικονομία. Επίσης εστιάζουμε ιδιαίτερα στην κατάρτιση. Συμφωνούμε όλοι σχετικά με τη σημασία των ψηφιακών προσόντων, σχετικά με, την κοινωνική, ε, με το κοινωνικό μη αποκλεισμό. Και δεν βλέπω να έχουν γίνει πολλά από την κατεύθυνση αυτή. Το σημείο το σημαντικό αφορά στις υποδομές. Χωρίς κατάλληλες ε, υποδομές ε, είναι περτό να ζητήσουμε τα υπόλοιπα. Η πρόσβαση στο διαδίκτυο είναι θεμελιώδες και θα πρέπει να υπάρξει ευρυζωνικό δίκτυο και στις ε, αγροτικές περιοχές και να καλύψει όλες τις οικογένειες. Τρίτη πτυχή αφορά τη συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Θα υποβάλουμε τροποποίησεις βελτιωτικές έτσι ώστε η ενιαία η αγορά δεν μπορεί να επιτευχθεί δίχως τη συμμετοχή των επιχειρηματιών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Με την ευκαιρία αυτής της μεικτής συνεδρίασης θα καλέσω όλους να μην χάσουν την ολιστική προσέγγιση. Εντάξει, ο καταμερισμός των αρμοδιοτήτων, αλλά θα είναι θεμελιώδες στο μέλλον η νομοθετική διαδικασία να είναι σύγχρονη με τους καιρούς. Ευχαριστώ. Επόμενος αγορτής, ο Φάρκο, Μάρκο Ζούλο από την ΙΜΚΟ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τις συζητήτριες για την εργασία τους και για την ισορροπημένη προσέγγιση που χρησιμοποίησαν. Δεν θα ήθελα να χάσουμε από το, στόχο μας με αυτή την πρώτη έκθεση μπορεί να θεωρηθεί ως εισαγωγική σε μια μακρά διαδικασία και προδιορίζουμε λοιπόν τον ορίζοντα στον οποίο θέλουμε να κατευθυνθούμε. Σε αυτόν τον ορίζοντα να μπορούμε να πούμε ότι η κοινωνία μετατρέπεται Άρδιν. Η ψηφιακή διάσταση πρώτα ήταν ένα μέσο, τώρα γίνει ένας τρόπος διαβίωσης των προσώπων. Σε αυτόν τον ορίζοντα λοιπόν βλέπουμε αυτό που μπορούμε να προσδιορίσουμε ως την, τον ψηφιακό η ψηφιακή υπηκότητα. Προκειμένου αυτή η, να οικοδομηθεί με τρόπο σταθερό, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε κάποιους πυλώνες. Πρώτα απ' όλα ο πυλώνας της ισότητας, διότι οι πολίτες, ε, οι χρήστες θα πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα, αλλά και τις ίδιες ευκαιρίες πρόσβασης στις υπηρεσίες και το περιεχόμενο και τα αγαθά. Ως εκ τούτου λοιπόν προβληματικές όπως ε, αυτό το geo-blocking ε, προκαλούν και αποτελούν διακρίσεις, διακριτική μεταχείριση. Ε, συμμετοχή η οποία θα πρέπει να είναι από πλευράς Χριστών ενεργός και ως εκ τούτου απαιτείται να ευνοήσουμε, να διευκολύνουμε την πρόσβαση της υπηρεσίας αφενός και αφετέρου να φροντίσουμε όλες τις δομές διακυβέρνησης αυτής της δυνατότητας πρόσβασης να είναι διάφανες. Τέλος, μια πιο εύκολη ανταλλαγή δεδομένων σημαίνει παράλληλα και μεγαλύτερο κίνδυνο για τους πολίτες. Δεν χρειάζεται λοιπόν οι πολίτες χρήστες να χάσουν την εμπιστοσύνη. Αλλά αυτό θα πρέπει να γίνει μέσω της προστασίας. Δεν πρέπει να είναι πραγματική, αλλά θα πρέπει να γίνεται ε, αντιληπτή. Δίχως την ε, εμπιστοσύνη και αξιοπιστία δεν μπορέσουν να ε, χρησιμοποιήσουμε τη δυναμικότητα αυτού του συστήματος. Αναφέρομαι στην πρακτική μετατροπής ε, των ε, προφοριών σε ένα μέσο εμπορίου ανάμεσα στα επιχειρήσεις. Αυτά τα δικαιώματα, τα ίδια δικαιώματα μάλλον σημαίνει να τροποποιήσουμε σε κάτι πιο πρακτικό τις δυνατότητες ε, του πολίτη. Χρειάζεται λοιπόν οι λύσεις ε, να μην αποτελούν μόνο με τις εναρμόνισεις του δικαίου. Συνοψίζονται λοιπόν ισότητα, συμμετοχή και εμπιστοσύνη είναι οι πυλώνες ε, για να οικοδομήσουμε την μελλοντική ψηφιακή υπηκότητα ή ηθαγένεια. Ευχαριστώ κυρία Κάπολ, έχει το λόγο από τη DNF. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τις δύο εισηγήτριες και για τη στρατηγική αυτή τη ενιαία εσωτερική ψηφιακή αγορά στην Ευρώπη, που είναι ένα πολύ περίπλοκο σύνθετο έγγραφο και πολλές κοινοβουλευτικές επιτροπές ε, έχουν τις δικές τους ξεχωριστές απόψεις που πρέπει να εξεταστούν. Απαιτούνται πολλά πράγματα και είναι πολύ καλή δουλειά που έχει γίνει. Ουσιαστικά αναφέρθηκαν τα τρία στοιχεία ε, που σε αυτό το στρατηγικό έγγραφο της Επιτροπής για την Ψηφιακή Ευρώπη προτείνονται, έχουν ληφθεί υπόψη και είναι πολύ ενδιαφέρουσα η καλύτερη προσπελασιμότητα για το διαδίκτυο, αναφέρθηκε ήδη, είναι ένα από τα προαπαιτούμενα. Είναι ένα μεγάλο δυναμικό σε αυτό το έγγραφο. 7 δις ευρώ εξοικονόμηση για τους Ευρωπαίους καταναλωτές αν μπορέσει να διαμορφωθεί με βελτιωμένα πλαίσια αυτή η αγορά. Μεγάλο ποσοστό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτήν την αγορά και έτσι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα μπορούν και οι startups να ε, δραστηριοποιηθούν δημιουργία προϋποθέσεων για νέα σύγχρονα δίκτυα και καινοτόμα δράση. Είναι σημαντικό αυτό, διότι οι μεγάλοι όγκοι δεδομένων πρέπει να μπορούν να καλύπτονται και να ρυθμίζονται. Στο νομοθετικό πεδίο και του ε, ΦΠΑ, ΦΠΑ και το δίκαιο του ανταγωνισμού πρέπει να λαμβάνεται υπόψη με ελέγχους και στον ψηφιακό τομέα. Όλα αυτά είναι καινούργιοι νέοι τομείς που ο ψηφιακός κόσμος δημιουργεί και χρειαζόμαστε νομικά πλαίσια για όλα αυτά. Και μέσα στο πλαίσιο αυτό φυσικά την ενίσχυση των καταναλωτών ώστε να έχουν εμπιστοσύνη στους παρόχους και τα προϊόντα στην ψηφιακή αγορά που θα προσφέρονται. Θέλω να αναφερθώ στην βέλτιστη χρήση του ε, δυναμικού ανάπτυξης. Ε, έχουμε υπόψη ότι η διεύρυνση, η επέκταση της ψηφιακής αγοράς θα δώσει 450 δις ευρώ επιπρόσθετα στην Ευρώπη. Αυτό ουσιαστικά αυτά προέρχονται μέχρι σήμερα από παραδοσιακούς επιχειρησιακούς κύκλους και δραστηριότητες και όχι τόσο από τον ε, ψηφιακό κόσμο και πρέπει να δούμε και το υπολογιστικό νέφος ε, το cloud computing όλα αυτά τα πλαίσια πρέπει να βελτιωθούν και όταν θα έχουμε 50 ε, δις τα οποία θα μπορούν να εξοικονομηθούν με αυτή την ψηφιοποίηση, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Η δική μας Κοινοβουλευτική Επιτροπή είχε δραστηριοποιηθεί και είχε συνεισφέρει σημαντικά προς αυτές τις προτάσεις. Ένας πολύ σημαντικός τομέας είναι εκείνος ο οποίος αφορά την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στην Ευρώπη. Μέχρι το 2020 με την ανάπτυξη της, ευ, ζώνη ε, του, της ε, ζώνης, του ευρυζωνικού φάσματος, είναι πολύ σημαντική υπόθεση. Καινοτόμες δηλαδή ρυθμίσεις που θα, δώσουν ένα πλαίσιο καλύτερου ανταγωνισμού. Χρειαζόμαστε και νέα, δεξιότητε νέες δεξιότητες από τους πραγματογνώμονες, ώστε ο τομέας αυτός να μπορεί να αναπτυχθεί όπως πρέπει. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κυρία μου. Σωστά αναφέρατε ότι σχεδόν 10 κοινοβουλευτικές επιτροπές που εμπλέκονται σε αυτό το κοινοβούλιο αναζητούν τις σωστότερες απαντήσεις σε σχέση με τις προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής. <clears throat> από πλευράς της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τον Αντιπρόεδρό της και με πολλούς επιτρόπους που συνεμπλέκονται εργάζεται σκληρά, εργάζονται όλοι αυτοί έντονα για να προαχθεί αυτό το θέμα. Και γύρω από αυτήν ε, όλη τη διεργασία πρέπει να σας πω ότι έχουμε και επισκέπτες που καλωσορίζουμε στο Ευρωκοινοβούλιο και έχουμε επίσης έχουμε δύο κοινοβουλευτικέ επιτροπές τη εσωτερική ε, αγοράς και των δικαιωμάτων των καταναλωτών και ε, της βιομηχανίας, τη έρευνας ε, και ενέργειας. Και έχουμε 120 μέλη ευρωβουλευτέ συνολικά από κοινού, κάθονται στις μπροστινές γραμμές και έχουμε μετά τους βοηθούς, συμβούλους, πολιτικούς συμβόλους, εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Συμβουλίου, οι συζητήσεις γίνονται μεταξύ των μελών, των μελών των δύο κοινοβουλευτικών επιτροπών μας εδώ. Και προσπαθούμε στις συζητήσεις μας να αντιμετωπίσουμε και να εξετάσουμε πολύ σημαντικά θέματα της ενιαίας ψηφιακής αγοράς. Θα ήθελα να δώσω τώρα την προεδρία στη συμπρόεδρο, κυρία Βίκη Φόρντ, της Επιτροπής ΣΥΜΚΟ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Για το διοργανωτικό τμήμα που έχεις εσύ που ξέρεις ποιοι θα μιλήσουν και εγώ αναλαμβάνω εκείνο το τμήμα το οποίο πρέπει να μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε το χάος γιατί όλοι θα θέλουν να παρέμβουν. Θα σας πω ποιοι είναι στον πίνακα αγοριτών μέχρι τώρα και στο συγγνώμη αν ξέχασα κάποιον. Να σηκώσετε το χέρι να μου το θυμηθείτε. Ah, Verheyen, Schaffhauser and Michael boni who is also the Libe rapporteur. Who else would like to be... Ποιος άλλος θα θέλει να πάρει το λόγο να προσθεθεί στο κατάλογο μελητών. Παρακαλώ, κάντε μου ένα σήμα. You didn't? Yeah, Okay. One, I don't know how that. That's okay. It's okay. It's just a. Sorry, sorry, Pilar, you will be on the list. Ναι, Pilar, μην ανησυχείς. Θα είσαι στον κατάλογο. Oh, you took. Because there were so many people. Όχι, απλώς δεν ήξερα πώς λειτουργούσε το σύστημα. Εντάξει. Προσθέτω και την Pilar. Mr. Zander. And who's the person in... Okay. Λοιπόν, θα προσπαθήσω κάπως να τα αναμίξω τα πράγματα μεταξύ των ε, δύο επιτροπών και των πολιτικών ομάδων, για να υπάρχει κάποια ισορροπία. Πριν ε, ξεκινήσω οποιοδήποτε άλλο, θα δώσω το λόγο στον εισηγητή της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ, τον κύριο Μπόνι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τις δύο εισηγήτριες. Νομίζω ότι έκαναν εξαιρετική δουλειά. Είναι μια πολύ καλή έκθεση. Και νομίζω ότι θα παραμείνει εξαιρετική μέχρι το τέλος. Θεωρώ ότι χρειαζόμαστε λύσεις που θα δημιουργήσουν και θα διαμορφώσουν ένα πλαίσιο εναρμόνισης μεταξύ διαφόρων τομέων και κλάδων, αλλά και κρατών μελών. Αυτός είναι ο κύριος στόχος της ενιαίας ψηφιακής στρατηγικής, να εναρμονίσουμε και να έχουμε μία λύση και όχι 28 διαφορετικά συστήματα, σε κάποιους τομείς βεβαίως, ε, τους οποίους θα πρέπει να εντοπίσουμε εμείς, αυτό είναι το καθήκον μας. Δεύτερον, χρειαζόμαστε λύσεις που θα συνεχίσουν να καλύπτουν την πραγματικότητα και στο μέλλον. Πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε και την νομοθεσία αλλά και την τεχνολογία και να κατανοήσουμε ότι η τεχνολογία κινείται ταχύτερα. Επομένως, χρειαζόμαστε ισχυρές νομοθετικές ρυθμίσεις, αλλά σε κάποιους τομείς χρειαζόμαστε και το λεγόμενο soft law και μη νομοθετική δραστηριότητα δηλαδή. Γιατί αυτό είναι καλύτερο για την ε, ψηφιακή εξέλιξη της Ευρώπης. Και το τρίτο σημείο που ήθελα να αναφέρω που συνδέεται με τη ΛΥΜΠΕ, σε αυτόν τον νέο τομέα, ή μάλλον σε αυτή την νέα εποχή, χρειαζόμαστε λύσεις που θα είναι αξιόπιστες. Πολύ σημαντικό αυτό το στοιχείο. Στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ ξεκινήσαμε τις εργασίες μας και θα γίνει συζήτηση στην Επιτροπή μας. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι πρέπει να υπάρξει συμμόρφωση με όλες τις πρωτοβουλίες που διαμορφώνονται υπό τη στρατηγική, την είναι ψηφιακή στρατηγική. Βεβαίως και η προστασία δεδομένων θα πρέπει ε, να συνδυάζεται με ισορροπημένο τρόπο με τις επιχειρηματικές δυνατότητες και την οικονομική ανάπτυξη. Πρέπει λοιπόν να βρούμε αυτή την κατάλληλη ισορροπία μεταξύ της προστασίας δεδομένων που είναι θεμελιώδες δικαίωμα και των επιχειρηματικών και οικονομικών ευκαιριών. Αυτό είναι ένας ε, βασικός ε, στόχος μας στι συζητήσει στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Επίσης, πρέπει να κατανοήσουμε και την σκοτεινή πλευρά του διαδικτύου. Η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ θα επικεντρωθεί στην καταπολέμηση του παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο και ε, θα αντιμετωπίσει και το ζήτημα του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο. Χρειαζόμαστε λοιπόν καλύτερου κανόνε ασφαλεία και μια εναρμονισμένη ανταπόκριση, αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε πολλούς τομείς που αυτή τη στιγμή δεν είναι ασφαλής. Και πρέπει να συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση για τα όσα συμβαίνουν ε, και στο πλαίσιο της ε, σχετικής οδηγίας. Ε, συγγνώμη, πρέπει να σε διακόψω. Α, τελευταίο σημείο. Ψηφιακή οικονομία. Δεν θέλουμε να επικεντρωθούμε μόνο στην προστασία δεδομένων αλλά και στο σύστημα της ιδιοκτησίας των δεδομένων. Γιατί θέλουμε μια οικονομία με οδηγό τα δεδομένα και νομίζω ότι θα υπάρξει συνεργασία μεταξύ όλων των επιτροπών για αυτό το θέμα. Σα έδωσα ένα λεπτό παραπάνω, γιατί μιλήσατε και εξ ονόματο τη Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Αλλά γενικά θα πρέπει να ε, κρατήσουμε το χρονικό όριο. Η Πίλαρ Sorry, I will ε, speak in, ε, Θα μιλήσω Πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια στις δύο συνεισηγήτριες, γιατί δεν είναι καθόλου εύκολο το έργο αυτό. Και κατάθεσαν ένα έγγραφο το οποίο θα είναι εξαιρετική βάση εργασίας για να αναπτύξουμε το έργο μας υστερότερα, μεταγενέστερα. Είναι σημαντικό να έχουμε ένα όραμα συνολικό για την κατάσταση που έχουμε μπροστά μας και πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Αν πρέπει να έχουμε κατακαιρματισμένες προτάσεις ε, νομοθετικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση στα ψηφιακά όπως και αλλού, είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την ευθύνη μας, να πάψουν να υπάρχουν φραγμοί και όρια μεταξύ κοινοβουλευτικών επιτροπών, μεταξύ τέτοιων σημαντικών θεμάτων, όταν γνωμοδοτούμε για αυτά τα θέματα. Πρέπει να καταβάλουμε κοινή προσπάθεια για να δώσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και είμαστε ικανοί να δώσουμε, για να προαγάγουμε το καλύτερο περιβάλλον ως πλαίσιο, για να μπορέσει να προαχθεί η ενιαία εσωτερική ψηφιακή αγορά είναι κάτι που έχουμε ως καθήκον να κάνουμε και πρέπει να δεσμευτούμε. Τρία πράγματα θέλω να τονίσω που είναι πολύ σημαντικά και πρέπει μόνιμα να λαμβάνουμε υπόψη. Δεν υπάρχει αντίφαση μεταξύ καινοτομία, μεταξύ ανταγωνισμού και μεταξύ του γεγονότος ότι πρέπει να αναπτυχθούν δίκτυα νέας γενεάς που χρειάζονται νέα, ε, νέα συνδρομή και νέες υποδομές που είναι απόλυτες αναγκαίες προϋποθέσεις. Δεν υπάρχει μια τέτοια αντίφαση. Είναι το πρώτο στερεότυπο που πρέπει να ε, σπάσουμε. Για την ψηφιακή αυτή αγορά πρέπει να υπάρχουν ίσες ε, προϋποθέσεις και όροι για υπηρεσίες που θα προσφέρονται με νέους κανόνες Πρέπει να έχουμε την αρχή της ισότητας. Αν ένας έχει παρόμοια η ίδια ε, υπηρεσία που παρέχει με κάποιον άλλο, πρέπει ισότιμα με τον ίδιο τρόπο να αντιμετωπίζεται. Όχι να ρυθμίζεται περισσότερο από ό,τι πριν, αλλά με ίδιο και ίσο τρόπο, δίκαια. Και η διαλειτουργικότητα είναι θεμελιώδου σημασία ώστε οι χρήστε να έχουν εναλλακτικέ λύσει στη διάθεσή του και να μην εξαρτώνται μόνο από έναν πάροχο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι είναι μια ιστορική στιγμή που είμαστε όλοι στον ίδιο χώρο και είναι πολύ σημαντικό, όπως ανέφερε και η Πιλάρ, να ενεργήσουμε από κοινού για να διαμορφώσουμε μια πραγματικά ενιαία ψηφιακή αγορά. Κάποιε κύριε παρατηρήσει, βέβαια κάποια έχουν ήδη υποθεί, το θέμα τη προσβασιμότητα, ευρυζωνικό δίκτυο, βασικά πρότυπα και είναι σημαντικό που είμαστε όλοι εδώ. Δεν εξετάζει κανεί σε βάθο τι δεξιότητε και πόσο σημαντικό αυτό το στοιχείο για να είναι και οι πολίτε μα έτοιμοι και σήμερα αλλά και στο μέλλον και πώς θα διαμορφώσουμε το ε, κατάλληλο σχολικό πρόγραμμα, αν θέλετε, για να είναι ε, όλοι οι πολίτες μας έτοιμοι. Ο γιος μου, έχω ένα γιο 9 χρονών, ήδη ε, ξέρει να χρησιμοποιεί όλες αυτές τις νέες τεχνολογίες και αυτό πρέπει να συνεχιστεί και στο μέλλον. Και βεβαίως τέλος η νοοτροπία. Πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη σε αυτή την ψηφιακή επανάσταση που όλοι βιώνουμε. Είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου αυτή τη στιγμή και θα έχουμε τεράστιες προκλήσεις. Αλλά αν τα πάμε καλά και σε αυτό το κοινοβούλιο, τότε και οι επόμενες γενιές θα μας ευχαριστούν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, μου δώσατε τη δυνατότητα να πω δύο λόγια. Και ελπίζω έτσι να ξεκινήσει και ένας διάλογος. Γιατί έχει επικρατήσει σιωπή στις επιτροπές μας. Επομένως, είναι καλό και πολύ θετικό να γίνεται αυτή η συζήτηση μεταξύ των επιτροπών. Άντρες Σουάπ. Ο κύριος Σουάπ, ευχαριστώ πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, με όλη την αισιοδοξία για αυτό το θέμα, δύο παρατηρήσεις θέλω να αναφέρω που θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικές. Το θέμα της ενιοποίησης των όρων για την πρόσβαση στην αγορά και των νομικών διατάξεων είναι ένα θέμα που στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εδώ και χρόνια μας απασχολεί και επανειλημμένα διαπιστώσαμε ότι στο τέλος είναι πάρα πολύ δύσκολη αυτή η ενιοποίηση, αυτό το ενιαίο νομικό πλαίσιο ώστε να επιτύχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Αν δεν πετύχουμε όμως την ενιαία εσωτερική αγορά δεν θα λειτουργήσει αυτή η ψηφιακή αγορά τα εμπόδια όμως τα οποία έχουμε μπροστά μας, αν έχουμε μια διαφορετική κατάσταση μεταξύ 28 κρατών μελών, είναι τεράστια τα εμπόδια αυτά. Και θα τα καταφέρουμε μόνο αν από κοινού μεριμνήσουμε και διοργανώσουμε τα πράγματα ώστε σε ένα ενιαίο πλαίσιο να καταλήξουμε πανενοσιακά η κυρία Κάλλας μίλησε για το δυναμικό και τη χρήση αυτού του δυναμικού. Αυτό όλο και περισσότερο με την αγγλική γλώσσα είναι κάτι το οποίο απλουστεύει τα πράγματα. Αλλά για μια πραγματική ενιαία εσωτερική αγορά στην Ευρώπη η γλωσσική φραγμή, τα γλωσσικά εμπόδια εξακολουθούν να υφίστανται και με όλη την αισιοδοξία δεν πρόκειται να καταργηθούν τα επόμενα δύο χρόνια. Επίσης στο ΦΠΑ έχουμε μια παρόμοια κατάσταση. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις λένε ότι υπάρχουν διεθνείς κανονισμοί και ρυθμίσεις που είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστούν από αυτές. Και όσον αφορά το geo-blocking, πολλές συζητήσεις θα έχουμε φυσικά επ' αυτού. Ένα θέμα είναι σημαντικό. Να δούμε πού θα υπάρχουν διακρίσεις όταν θα υπάρχουν νομικά ε, τα επιχειρήματα για ε, τις διαφορές μεταξύ των κρατών μελών και φοβούμε θα υπάρξουν μια ολόκληρη σειρά τέτοιων ε, εμποδίων. Ελπίζω όμως ότι θα τα καταφέρουμε να τα αντιμετωπίσουμε. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ένας ακόμα μιλητής από τους Σοσιαλδημοκράτες ε, και μετά ένας από ECR, άλλα και ΕΝΕΦ. Όλγα Σιναλόβα. Ευχαριστώ. Εφόσον υπάρχει και διερμηνία στην ε, τσεχική, θα μιλήσω τα τη μητρική μου γλώσσα. Ευχαριστώ που μου δώσατε τον λόγο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τις δύο ε, συντάκτριες ε, αυτών των εκθέσεων. Είναι εξαιρετικές ε, και αντιμετωπίζουν πολλά θέματα από πλευρά της προσέγγισης αυτής αλλά κάνουμε λόγο για τις αρχές τις βασικές θεμελιώδεις αρχές της αγοράς είτε είναι online είτε είναι offline Πρέπει να μιλήσουμε για την αξιοπιστία και τις δίκαιες αρχές που πρέπει να εφαρμόζονται, κυρίως για την αξιοπιστία και το κύρος τους. Και αυτό συναρτάται με τις αρμοδιότητες των εποπτικών οργάνων. Εδώ πάλι χρειαζόμαστε δυναμικό, επαρκές δυναμικό και επαρκείς αρμοδιότητες για να λειτουργήσουμε σωστά. Είναι πολύ σημαντικό να σκεφτούμε πώς θα προστατέψουμε τους καταναλωτές αλλά αυτό συσχετίζεται και με έναν άλλο τομέα. Κάνουμε λόγο φυσικά για δέσμες μέτρων, για πακέτα μέτρων και που ζητούμε συγκεκριμένες προτάσεις. Και αυτά δεν αφορούν μόνο αποκλειστικά τις τιμές, την τιμολόγηση αυτών των υπηρεσιών και ε, την αποστολή τους. Πρέπει να δούμε και το χρονικό διάστημα το οποίο τα πακέτα αυτά τα θέματα αυτά βρίσκονται καθοδόν όταν έχουν παραγγελθεί. Είναι πολύ σημαντικά αυτά τα θέματα για τους καταναλωτές που θέλουν να χρησιμοποιήσουν τέτοιες υπηρεσίες ε, αποστολής δεμάτων και αγαθών. Για τις υπηρεσίες ε, χαίρομαι για το ότι γίνεται λόγος για το geo-blocking, διότι το geo-blocking είναι ένα θέμα πάρα πολύ προβληματικό και δεν αφορά μόνο τη διάκριση αλλά και κριτήρια τιμών αλλά πρόκειται επίσης και για το θέμα της ελεύθερης πρόσβασης όλων των καταναλωτών σε ίδιες οι κοινές υπηρεσίες. Ευχαριστώ. Όσοι βρίσκονται στο κατάλογο μιλητών θα έχουν την δυνατότητα να μιλήσουν, μην ανησυχείτε. Dan Dolson, Robert Rosford, Schaffhausen. Γιατί από ό,τι κατάλαβα πρέπει να φύγει. Δεν ξέρω αν κάποιο πρέπει να φύγει πιο νωρί να μου το πει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ τις δύο εισηγήτριες. Ένα πολύ καλό πρωτοκείμενο. Πρέπει να αναγνωρίσουμε πρώτα απ' όλα ότι ήδη βρισκόμαστε στην ψηφιακή επανάσταση και αυτό θα αναταράξει τα νερά. Όμως το πιο σημαντικό είναι ότι θα ενδυναμώσει και τους ε, επιχειρηματίες και τους καταναλωτές. Πρέπει να είμαστε θετικά διακείμενοι και όχι αρνητικά. Είναι μια θετική εξέλιξη. Η εμπιστοσύνη είναι βεβαίως ε, σημείο κλειδί και επιχειρήσει. Είναι πολύ σημαντική η επιμερισμένη οικονομία. Ε, πρέπει να υπάρξει εμπιστοσύνη. Από οικονομική σκοπιά αυτό είναι τεράστιο όφελο. Από την ευεσμένη οικονομία βλέπουμε ότι οι καταναλωτέ και οι εργαζόμενοι δεν χρειάζονται απαραίτητα την υφιστάμενη νομοθεσία. Γι' αυτό θα πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Σε ό,τι αφορά τώρα συγκεκριμένε παρατηρήσει για την πρόταση, για, το γεωγραφικό αποκλεισμό, θεωρώ ότι ο δικαιολόγητο γεωγραφικό αποκλεισμό ε, είναι αρνητικό, για παράδειγμα στο κρίκετ στην Ισπανία ή οι γαλλικές ταινίες στη Σουηδία. Για μένα λοιπόν η φορητότητα του, ε, νομι... του νομίμως αποκτηθέντος περιεχομένου είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να διασφαλιστεί. Για το ηλεκτρονικό εμπόριο δεν νομίζω ότι χρειαζόμαστε νέα νομοθεσία. Τα επιγραμμικά εργαλεία εμπιστοσύνη νομίζω ότι επαρκούν και όπως ε, όλοι οι υπόλοιποι κλάδοι της βιομηχανίας πρέπει και εδώ με τα, τις υπηρεσίες αποστολής δεμάτων ε, θα πρέπει να ισχύσει το ίδιο. Για τις τηλεπικοινωνίες, συντονισμό, συνεργασία, αλλά δεν συμφωνώ με, την, ε, με τον αρμονισμένο φάσμα ούτε με τον υπάρξει ενιαία ρυθμιστική αρχή σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τέλο, να μην είμαστε υπερπροστατευτικοί, να μην υπάρχει δηλαδή προστατευτισμό. Δεν πρέπει να μπλοκάρουμε την Ευρώπη και να την κλείσουμε από όλη από όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Αναφέρθηκε προηγουμένω ότι το 54% του περιεχομένου προέρχεται από τη ΣΥΠΑ. Αυτό συμβαίνει γιατί παρέχουν ε, το προϊόν και τι υπηρεσίε που θέλουν οι καταναλωτέ. Εμεί εκεί δεν το κάνουμε. Πρέπει να εξετάσουμε ολόκληρο τον κόσμο, όχι μόνο του Ευρωπαίου καταναλωτέ. Ευχαριστώ. Ρόμπερτ Ευχαριστώ για τις δύο εισηγήτρες για την πολύ καλή έκθεση. Η επανάσταση ε, την οποία δρεχόμεθα είναι μια βαθιά επανάσταση βιομηχανική, η οποία όμως ε, αναταράζει τα πάντα. Τον τρόπο παραγωγής, τον τρόπο κατανάλωσης και τον τρόπο ζωής μας ακόμα. Πρέπει να δούμε το μέλλον. Και αυτή η έκθεση αυτό μα καλεί να κάνουμε, αλλά πρέπει να πάμε ακόμα παραπέρα. Είναι η επιθυμία μα, μάλλον οι ζωέ ε, των παιδιών και των επόμενων γενεών. Πρέπει η Ευρώπη να βρεθεί σε αυτό το ραντεβού, να διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο, να μην ε, σέρνεται πίσω από τις ΗΠΑ ή από την, την Ασία. Να είναι ενωμένη με τις ε, δυνάμεις της και τις αξίες της. Χρειαζόμαστε μια βαθιά ψηφιακή οικονομία με τις μικρές επιχειρήσει, αλλά και με τους γίγαντες ε, τη ψηφιακή εποχή που πρέπει να συμβάλλουν με όλα του τα μέσα στην υλοποίηση της ψηφιακή στρατηγική. Η εμπιστοσύνη στις ψηφιακές τεχνολογίες είναι κάτι θεμελιώδου σημασία, το ξέρουμε όλοι. Εμείς όμως στην ε, ΙΜΚΟ ε, που εξετάζουμε ιδιαίτερως ε, τις μικρές επιχειρήσεις πρέπει να υπενθυμίσω ότι το έλλειμμα σε ό,τι αφορά και η έλλειψη ψηφιακών γνώσεων είναι το, η βασική πρόκληση και πολύ φοβάμαι ότι θα υπάρξει καθυστέρηση σε αυτό το τομέα. Γι' αυτό θα πρέπει να το εξετάσουμε αυτό με μεγάλη προσοχή. Τέλος, η ψηφιακή τεχνολογία ε, οδηγεί στην επιμεριζόμενη οικονομία. Βεβαίω υπάρχουν τεράστιε δυνατότητε. Όμω, προσοχή, αυτέ οι εξέλιξει μπορούν να είναι πολύ θετικέ και πολύ αρνητικέ. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα νομικό πλαίσιο και στο κοινωνικό επίπεδο, αλλά και στη φορά την προστασία του καταναλωτή. Η επιμερισμένη οικονομία μπορεί ε, να αποτελέσει ένα πλαίσιο ανταλλαγής ε, μεταξύ ατόμων ε, σε ένα άτυπο και ανεπίσημο πλαίσιο ή ακόμα και ένα χαοτικό σύστημα συναλλαγών χωρίς καμία προστασία. Πρέπει λοιπόν να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Είναι ένα πολύ καλό θέμα και πολύ καλή δουλειά που έχει γίνει μέχρι τώρα. Κύριε Σαφάουζα, αγαπητοί συνάδελφοι, οι τεχνολογίες δεν είναι ουδέτερες. Διαμορφώνουν τον κόσμο. Διαδίδουν ε, σκέψεις και τρόπους ε, σκέψης είναι ένας ε, τρόπος επιβολής ε, της εξουσίας ε, και της οικονομικής δύναμης. Μπορούμε να αφήσουμε κάποιες επιχειρήσεις να μας διοικούν. Ή θέλουμε να διαφυλάξουμε ένα, κάποιον έλεγχο στο μέλλον μας. Πρώτον, σε ό,τι αφορά ε, τον υπερβολικό ανταγωνισμό. Δεν διευκολύνει τις υποδομές, τις επενδύσεις στις ε, υποδομές. Αυτό προκύπτει από μια έκθεση του Γαλλικού Κοινοβουλίου, αλλά και από την δική μου εμπειρία από όσους επενδύουν σε αυτές τις υποδομές. Γιατί πολύ συχνά οι πειρατές είναι αυτοί που επωφελούνται χαμηλών τιμών, ε, καταραίει η αγορά και μόνο αυτοί κερδίζουν. Επομένως πρέπει να το προσέξουμε αυτό. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά τον αθέμητο τώρα ανταγωνισμό. Οι ΙΠΑ προστατεύονται από τους ε, μεγάλους ε, παρόχους ε, περιεχομένου. Τι κάνει η Ευρώπη για να προστατεύσει τον εαυτό τους όπως κάνουν οι ΙΠΑ. Και τρίτον, δεν πρέπει να μας ξεφύγει και η εθνική διάσταση, γιατί είναι πολύ σημαντικό ζήτημα ασφάλειας, άμυνας, προστασίας δεδομένων. Και δεν γίνεται να αφήσουμε κατά μέρο αυτή την εθνική διάσταση. Αν την αφήσετε εκτός, θα κάνετε μεγάλο λάθος και δεν θα καταλήξετε πουθενά. Ευχαριστώ. Εντάξει, θα σας πω τη σειρά να δώσω το λόγο σε μερικά ακόμα μέλη της ΣΥΤΡΑ και μετά θα ε, με, τι κινούμε μεταξύ διαφόρων πολιτικών ομάδων. Ζάντερ Μούντι. Νεν, Κοράτσα Μπιλτ, Ντάντι, Θουν, Ιακονσάρι, Τσοσνέσκι, and then getting me in great trouble because it's the fight. Και μετά τα Τάβγολτα Πέλτς και αυτό ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολο γιατί είναι και αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου. Δεν ξέρω αν κάποιος άλλος θέλει να πάρει τον λόγο. Σάντερ. Κυρία Σάντερ, ευχαριστώ. Είχα ένα πρόβλημα με το μικρόφωνο. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τις δύο εισηγήτριες για την έκθεσή τους. Να πω ότι συμφωνώ με κάποια από τα όσα αναφέρθηκαν. Πράγματι, η σημερινή ψηφιοποίηση είναι ένα σημαντικό διακύβημα για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση, αλλά πάντα από κοινού και 28. Εγώ θα ήθελα να επανέλθω στο ζήτημα ε, των πλατφορμών και την κακή ρύθμιση θεωρώ. Σήμερα βλέπουμε ότι οι μικρές και μεσές επιχειρήσεις δεν έχουν καμία διαπραγματευτική ισχύ με αυτές τις πλατφόρμες σε ό,τι αφορά τους όρους και προϋποθέσεις ε, συμμετοχής τους ή πρόσβασης τους σε αυτές τις υπηρεσίες. Δεν υπάρχει κανένας έλεγχος ε, για τις ε, διακρίσεις ή για την μη αναφορά τους. Ήθελα να κάνω δύο προτάσεις. Πρώτον, να εξετάσουμε το ενδεχόμενο θέσπισης μιας ταχείας προσέγγισης και διαδικασίας μάλλον ε, επίλυσης διαφορών, γιατί σήμερα η διαδικασία είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα. Αν δείτε για παράδειγμα με την Google, μπορείτε να φανταστείτε ένα, θα μπορούσαμε να φανταστούμε ένα σύστημα πολύ πιο γρήγορο, όπως γίνεται στον ε, κλάδο των τηλεπικοινωνιών, για παράδειγμα. Δεύτερη πρόταση, εφαρμογή ενός, ε, ενός ε, οργανισμού βαθμολόγησης ε, και αξιολόγησης, ενός οίκου αξιολόγησης αν θέλετε, των πλατφορμών αυτό. Και αυτό θα μπορούσε να μας βοηθήσει ε, να διευκολύνουμε και τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές. Ευχαριστώ. Claire Moody. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τις εισηγήτριες για αυτή την έκθεση. Είναι μια εξαιρετική αρχή. Βεβαίως και έχουμε πράγματα να προσθέσουμε. Πρώτον, μεγάλη έμφαση δίνουμε στον καταναλωτή και αυτό είναι κατανοητό. Όμως η ενιαία ψηφιακή αγορά είναι κάτι πολύ ευρύτερο. Υπάρχει ένα πολύ ισχυρό στοιχείο business to business μεταξύ των επιχειρήσεων δηλαδή και αυτό θα πρέπει να αναγνωριστεί και εδώ. Δεύτερον, για τις υποδομές. Δίνεται έμφαση ε, στην διευκόλυνση των ε, ιδιωτικών επενδύσεων στις υποδομές. Όμως, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι υπάρχει και δημόσιος ρόλος σε τομείς που είναι πιο δύσκολο να προσελκύσουν ας πούμε, τις ιδιωτικές επενδύσεις. Αυτό μπορεί να αφορά την διεύρυνση του Wi-Fi, το σύνδεμα του δικτύου ή και βασικές υποδομές. Πρέπει να αναφερθεί και αυτό. Και τρίτον, οι πολίτες που είναι αποδέκτες όλων αυτών. Έχουμε για παράδειγμα την απασχόληση. Πρέπει να εξετάσουμε την επέκταση, τη διεύρυνση της επισφαλούς εργασίας και της ε, πλήρους απασχόλησης. Σε αυτό θα πρέπει να υπάρξει διαβούλευση με ε, κοινωνικούς εταίρους, εργοδότες, συνδικάτα, για να βρούμε κοινέ λύσεις για τη μορφή που θέλουμε να πάρει το μοντέλο απασχόλησης στο τέλος διαδικασίας. Και να υπάρξει μια εξισορρόπηση μεταξύ των όσων έχουν πρόσβαση σε ασφαλή δουλειά και σε όσους δεν έχουν. Και σε ό,τι αφορά την διαβίου μάθηση, πρέπει να είναι κάτι το οποίο θα ενισχυθεί. Δεν μπορεί κάποιο να έχει στο μυαλό του ότι η παιδεία που θα λάβει, η εκπαίδευσή του, α πούμε, σταματάει στα 18 ή στα 21 ή όποτε σταματάει ο καθένα. Και όλοι να έχουμε πρόσβαση στην ε, ψηφιακή συμπερίληψη μέσω τη διαβίου μάθηση. Άννα Μαρία Κρατσπίλτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και εγώ τις δύο συγγήτρες και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πολύ καλό αυτό σχέδιο έκθεσης γιατί έτσι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε καλύτερα από κοινού τι προκλήσει τη νέα ψηφιακή αγορά. Είναι μία έκθεση πλαίσιο, επομένω να θίξω κάποια κέρια για μένα ζητήματα. Πρώτον, μιλήσαμε για ένα διαδίκτυο που θα είναι δωρεάν, ανοιχτό, ελεύθερο μάλλον, ανοιχτό και παγκόσμιο. Όλα που αναφέρθηκαν αυτά για το ευρωπαϊκό υπολογιστικό νέφος και όλα την ψηφιακή ακαιρεότητα και το καθεξής, όλα αυτά θα πρέπει να βγουν δεν θα γίνουμε εξίσου ανταγωνιστικοί με το υπόλοιπο κόσμο αν αφήσουμε απ' έξω τους υπόλοιπους. Πρέπει να διαμορφώσουμε ένα ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού στην Ευρώπη, να ε, καταργήσουμε τους φραγμούς και τα εμπόδια και να απλοποιήσουμε τους δικούς μας κανόνες. Δεύτερον, η ψηφιακή επανάσταση είναι πολύ πιο γρήγορη ε, από ό,τι νομίζουμε. Και εμείς δεν έχουμε λάβει ακόμα τον ε, κύριο ηγετικό ρόλο. Πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό. Καινοτομία, τεχνολογία, επιχειρήσεις. Αυτή είναι στο, στη θέση του οδηγού. Δεν πρέπει λοιπόν να μείνουμε πίσω. Πρέπει να διευκολύνουμε με τον νομοθετικό μας ρόλο. Πρέπει λοιπόν σε αυτή τη διαδικασία, παρότι θα υπάρξει μια αναταρχή της αγοράς, ε, πρέπει να σταματήσουν, να σιωπήσουν επιτέλους τα εθνικά συμφέροντα. Και αυτός ο προστατευτισμός που ε, βλέπουμε σήμερα είναι η μεγαλύτερη απειλή στις νέες θέσεις απασχόλησης και την ψηφιακή αγορά. Κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Ασφάλεια δικαίου. Αυτό είναι ο δικό μου ρόλο και ε, με προβληματίζει ιδιαίτερω η απόφαση του δικαστηρίου ε, για το Safe Harbor. Ελπίζω η Κομισιόν σύντομα να δώσει κάποια ε, σαφήνεια και διευκρινήσει προ τι επιχειρήσει για το τι θα γίνει με τα δεδομένα. Και ταχύτατα θα πρέπει να υιοθετήσουμε τον κανονισμό για την προστασία δεδομένων με μια ε, προσέγγιση πιο φιλική προς τι επιχειρήσεις. Και καθώ και εγώ είμαι επιχειρηματία, σε ό,τι αφορά το ηλεκτρονικό εμπόριο, θα πρέπει να ανοίξει η αγορά για την παράδοση δεμάτων στην Ευρώπη. Μια καθολική προσέγγιση χρειαζόμαστε προ τι υπηρεσίε πολύ περισσότερο από ό,τι τώρα και κάποια στιγμή θα πρέπει να δούμε και το σύστημα Απλούστευση του ΦΠΑ. Ευχαριστώ. Νίκολα Ντάντι. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ και τις δύο εισηγήτριες ε, για τις πολύ καλές εκθέσεις. Θα ήθελα καταρχήν να ασχοληθώ με μια οριζόντια προσέγγιση του ζητήματος. Ε, το βλέπουμε για αυτήν τη συνεδρίαση αυτή μας ε, διαδεξάγεται εντό τη αίθουσα ονομέλεια για πρώτη φορά ίσως σημαίνει ότι προσεγγίζουμε την, ε, ε, ε, την ψηφιακή επανάσταση με τρόπο συνολικό. Αυτό έχει σημασία διότι καθημερινά ανακαλύπτουμε την ψηφιακή επανάσταση μόνο ότι δεν το αντιλαμβανόμεθα. Κατά τη γνώμη μου λοιπόν αυτό αποτελεί ένα από τα στοιχεία επαναπρόθεσης της ευρωπαϊκής οικονομίας. Δεν πρόκειται να επισέλθουμε εδώ σε λεπτομέρειες για όλες τις πτυχές της ε, ψηφιακής οικονομίας και της ε, old economy. Δηλαδή πώς θα μπορέσουν να δημιουργήσουν ευκαιρίες για τις νεοφυείς επιχειρήσεις. Όπως επίσης, ε, και το λέω ως μέλος της Επιτροπής Ιστορικής Αγοράς, το ίδιο το γεγονός ότι η ψηφιακή οικονομία ε, θα προχωρήσει χωρίς σύνορα, αυτό είναι πολύ σημαντικό για την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς. Και να κάνω τρεις ε, αναφορές. Ένα από τα βασικά στοιχεία θα είναι αυτό της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, η δυνατότητα να έχουμε διοίκηση ε, ψηφιακή. Αυτό σημαίνει ότι μειώνεται η γραφειοκρατία και έχουμε, απελευθερώνουμε διαφόρους πόρους. Κάτι ακόμα το οποίο θα πρέπει να είναι ασφαλές είναι ότι Χρειάζεται να επανακτήσουμε την ε, αξιοπιστία και την εμπιστοσύνη των πολιτών. Και οι πολίτες να γνωρίζουν ότι έχουν ένα δίκτυο ασφαλές, ε, σίγουρο, ε, για τις δραστηριότητε που γίνονται σε αυτό. Τώρα το ζήτημα της, του επιμερισμού της οικονομίας, δηλαδή μια οικονομία την οποία πετύχαμε χάρη στην ψηφιακή οικονομία, μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε με τρόπους διαφορετικούς από ότι την παλιά οικονομία, την old economy. Περιμένουμε εδώ ε, σημαντική συμμετοχή του Ευρωπαϊκής Επιτροπή ε, και εμείς θα συμβάλλουμε φυσικά για την επίτευξη αυτής, τη της ε, ανακοίνωσης. Ευχαριστώ. Επόμενη αγορήτρια. Ευχαριστώ. Ομολογώ πως εντυπωσιάζομαι από την συνεδρίαση που διεξήχθη πριν ακριβώ αυτή τη συνάντηση για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει και για το επιγραμμικό εμπόριο. Θα ήθελα να ασχοληθώ με αυτό το θέμα αφού ακούσαμε του περισσότερου από του συναδέλφου, όχι όλου. διότι πολλοί έκαναν παράπονα, έκαναν πάρα πολλέ ε, ερωτήσει και μετά έφυγαν από την αίθουσα. Θα ήθελα να επικεντρωθώ σε αυτό, το ζήτημα του e-trade, του ηλεκτρονικού εμπορίου. Κάποια ζητήματα με κατέθλιψαν. ε, χρόνια στο Κοινοβούλιο και συνεχίζουμε να μιλάμε για τα ίδια πράγματα. Θυμάμαι την πρώτη το φόρουμ για την ενιαία αγορά που διεξήχθη σε αυτήν εδώ την το 2005 κάπου, κάπου εκεί, το 2009 ίσως και ορισμένοι από εσά ίσως να ενθυμίσετε ότι ε, είδαμε μια σύντομη ταινία για, με το επιγραμμικό εμπόριο και θυμάμαι ότι υπήρξαν διάφορες μικρές ταινιούλες ε, που, που παρουσίαζε ε, μια αυστριακή έμπορο η οποία δεν μπορούσε να πουλήσει τα λάδια της ε, στην Γερμανία την Ιταλία διότι οι ταχυδρομικές υπηρεσίες κόστησαν τόσο πολύ και αυξανόταν αυτό το κόστος από τη που το προϊόν διέσυζε τα σύνορα. Θυμάμαι αυτή τη γυναίκα που έλεγε ότι έπρεπε ήθελε να αγοράσει κάποια ρούχα αλλά δεν ε, μπορούσε να το πράξει διότι υπήρχαν διάφορα εμπόδια τελωνιακής φύσης. Λοιπόν, σήμερα αυτές τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις άκουσα με ιδιαίτερη ενόχληση ομολογουμένως πάνω κάτω τα προβλήματα και ομολογώ ότι αυτό είναι ντροπή για όλους μας. Τώρα εργομίζομαστε σε μια έκθεση ιδίας πρωτοβουλία, αλλά αυτή η έκθεση ιδίας πρωτοβουλία, το γεγονό ότι επικεντρωνόμεθα στην εσωτερική ενία ψηφιακή αγορά, θα αποφέρει κάποιες συγκεκριμένες δράσεις. Ένα πρόγραμμα δράσης για, ε, για την παράδοση, για την ηλεκτρονική παράδοση. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα σαφή στόχο. Χρειαζόμαστε ονόματα των υπευθύνων. Και το άλλο το οποίο ελπίζω να πετύχουμε πρόοδο, ε, μια δράση για με ένα σαφή στόχο για την κατάργηση αυτών των 28 συστημάτων ΦΠΑ. Συμφωνώ με τον Φιλίπ και ολοκληρώνω. Εάν κάποιος πει ότι ε, ασχολούμεθα μόνο με τις ρυθμίσεις, ε, όχι δεν είναι γεγονό, δεν χρειαζόμαστε πολλές ρυθμίσεις, χρειαζόμαστε μία ενία. Ευχαριστώ. με Μέτση έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Συγχαρητήρια στις συγγήτριες, έκαναν πολύ καλή δουλειά και ε, ε, έθεσαν τις βάσεις για περαιτέρω συζητήσει. Τρία σημεία. Δεν θα χρειαστώ πολύ χρόνο. Προστασία των καταναλωτών, των δικαιωμάτων των και συγχαρών των καταναλωτών στην Ευρώπη είναι πολύ σημαντικό. Θα πρέπει να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών διαφορετικά δεν θα μπορέσει να προχωρήσει αυτή η ψηφιακή αυτό το ψηφιακή ψηφιακός αιώνας ψηφιακή εποχή η βάση όλων είναι η εμπιστοσύνη θα πρέπει να έχουμε κατά νου την ε, έκθεση του DCJ που μιλάει για το safe harbor regime για το καθεστώς ασφαλούς λιμένα Μελλοντικά μέτρα λοιπόν θα πρέπει να εγγυώνται υψηλό επίπεδο προστασίας. Δεύτερο σημείο που θα ήθελα να θίξω αφορά το πακέτο τηλεπικοινωνιών. Στο πλαίσιο των τριμερούς διαλόγου ε, δεν, ε, δεν ε, δεν πετύχαμε συμβασμούς ε, ιδιαίτερους ως Ήμικο. σχετικά με την οδηγία τα καθολικά δικαιώματα. Και αυτά τα ζητήματα λοιπόν θα πρέπει να εξεταστούν ε, συνεπώς, με τρόπο συνεκτικό, μια πλήρη μεταρρύθμιση είναι απαραίτητη. Τέλος, κάτι ιδιαίτερο σημαντικό, δεν μπορούμε να μιλάμε για ψηφιοποίηση εκτός εάν ασχοληθείτε και με το ζήτημα της ε, εκτύπωσης. Αυτά είναι τα τρία σημεία λοιπόν. Να σας ενημερώσω πως χρειάζεται να αναθεωρήσουμε την οδηγία για τις καθολικές υπηρεσίες και το θέμα των προστασίας των καταναλωτών που έθιξα και εγώ και ο κ. Μπούσακ μετά από τις αντίσεις που είχαμε τους επιτρόπους ε, την περασμένη εβδομάδα σχετικά με το πρόγραμμα του προσεχούς έτους. Ε, υπενθυμίζουμε λοιπόν αυτήν τη δέσμευση προκειμένου οι ε, διάφορες διαδικασίες να αναθεωρηθούν. Αγία Κασάρη, ευχαριστώ. Πολύ ενδιαφέρουσα, ενδιαφέροντα όλα αυτά. Χρειάζεται να είμαστε λίγο πιο ταπεινοί ενώπιον αυτής της ε, ψηφιακής εποχής μπορούμε να δεχθούμε ότι πρόκειται για ένα νέο ανεξερεύνητο έδαφος όπου υπάρχουν πολλές, πολλοί άγνωστοι η Επιτροπή λοιπόν θα πρέπει να ανελάβει την μελέτη που αφορά το τομέα της ψηφιοποίησης της ευρωπαϊκής κοινωνίας και των πολιτών. Θα πρέπει να εστιάζουμε σε κάποια όρους κλειδί. Συμμετοχή, πλήρης πρόσβαση, πλήρη συμμετοχή και ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες προσώπων που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες όπως ηλικιωμένοι και άτομα με αναπηρία που έχουν συμβάλει για πάρα πολλά χρόνια στην ευημερία μας και τώρα κινδυνεύουμε να αποκλείσουμε αυτά τα πρόσωπα και αυτό θα ήταν καταστροφικό. Ορισμένοι ανέφεραν τον όρο εμπιστοσύνη και μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Κάνουμε ελέγχους στα αυτοκίνητα για την οδική ασφάλεια. Θα πρέπει να ε, υπάρχουν αυτά τα προγράμματα και για τα συστήματα software. Είμαι βέβαιη πως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ηγηθεί αυτή της ε, προσέγγισης ζητήματα ασφαλείας. Ευχαριστώ, κυρία Φασινόφσκη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η ανάπτυξη των μέσων επικοινωνία και η επιτάχυση αυτών αποτελεί μια τάχιστη ε, ε, προσαρμογή των επιχειρήσεων. Γι' αυτό λοιπόν ε, οι επιχειρήσεις διαλαμβάνουν πολύ σημαντικό ρόλο και θα πρέπει να ευνοηθεί η επιστροφή σε μετά από την άγνωση των θέσεων της Κομισιόν μας αφήνει με πολλές εμβολίες. Μιλάμε εδώ για το μέλλον της Ευρώπης που αξίζει πολλά περισσότερα παρά παροχημένες ε, μελέτες που βλέπουμε σήμερα στις τραγικές συνέπειες η ολοκλήρωση της ε, ψηφιακής αγοράς αφορά τα οικονομικά συμφέροντα του συνόλου της Ένωσης. Αυτή η ομοσπονδιοποίηση οδήγησε σε μια απορρίθμιση των αγορών και των κεφαλαίων η οικονομική ανασφάλεια που έθιξε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά και τις μεγάλες καθώς επίσης και η απειλή της ε, ατομικές ελευθερίες. Θεωρώ θα πρέπει να δημιουργηθεί ε, ένα ε, κατάλληλο ευρωπαϊκό habitat. Μιλάτε για υποδομές και για κάλυψη, αλλά ποτέ για κόστος. Στη Γαλλία πολλές περιφέρειες δεν έχουν ακόμα 3G και εσείς συζητάτε το 5G τη σχέση έχει σε έξι που αναφέρει ότι μας απασχολούν διάφορες εθνικές προσεγγίσεις. και τι σημαίνει ε, ενεργό καταναλωτή στο πλαίσιο των ε, μικρών επιχειρήσεων. Εμεί λέμε ναι στην ψηφιοποίηση, ναι στην προστασία των καταναλωτών, ναι στην αποτελεσματική ε, πρόσβαση στι υπηρεσίε, ναι στην ανάπτυξη διοντολογία, αλλά όχι στα ομοσπονδιακά συμφέροντα που ο κ. Ζουβάμος ε, αποχώρησε, δεν πρέπει να σιωπήσουμε τα ε, εθνικά συμφέροντα. Η Ευρώπη περνάει μέσα από τα εθνικά συμφέροντα και όχι από την κατάργησή τους. Εμείς θα φροντίσουμε να τροποποιήσουμε όλες τις πτυχές αυτής της έκθεσης, καθώς επίσης και όλα όσα θα θεωρήσουμε ανεπαρκή για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των επιχειρήσεων και των καταναλωτών. Ευχαριστώ. Οι ε, συνάδελφοι Έργα Χόπνα και λοιπά είναι οι τελευταίοι τέσσερις αγορητές. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ζήτω συγγνώμη για την καθυστέρηση. Έπρεπε όμως να παρακολουθήσω μια άλλη συνεδρίαση και έπρεπε να βιαστώ να έρθω σε αυτή τη συνεδρίαση εδώ ανάμεσά σας. Θέλω να εκφράσω σε σχέση με το θέμα αυτό την αισιοδοξία μου. Όμως πέρα από αυτή την θετική αντιμετώπιση θεωρώ ότι πολλά πρέπει να γίνουν. Πολλά εμπόδια υπάρχουν ακόμα τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν. Και δεν μπορούμε να είμαστε αρκετά επιτυχείς αν δεν αντιμετωπίσουμε αυτά τα εμπόδια. Συζητήσαμε το θέμα διαμακρών και ελπίζαμε διαμακρών ότι θα μπορούσαμε να καταλήξουμε στην ψηφιακή εποχή. Είδαμε όμως ότι δεν είναι καθόλου τόσο εύκολα τα πράγματα. Αν δει κανείς το τι γίνεται στη ΣΥΠΑ, στις 66 από 100 εταιρείε που είναι ανταγωνιστικές σε αυτόν τον τομέα, 66% δεν ισχύει το ίδιο όμως δυστυχώς για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Δυστυχώς. Πολλά πρέπει να γίνουν και πρέπει να θέσουμε ενώπιόν μας αυτούς τους στόχους ώστε να είμαστε αποτελεσματικοί. Πολύ νομοθετικό έργο πρέπει να καλυφθεί. Να μπορούμε να υποστηρίξουμε αυτή την έκθεση και τις συνεισηγήτριες με απλά πράγματα ξεκινώντας, μειώνοντας, αντιμετωπίζοντας τα προσκόμματα σε σημαντικό βαθμό. Από την άλλη βέβαια πλευρά πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη ότι πρέπει να υιοθετήσουμε θετικά μέτρα στη συνδρομή μας αυτή, στην υποστήριξη των επιχειρήσεών μας όπου δεν είναι έτοιμες ακόμα να είναι ανταγωνιστικές σε αυτόν τον τομέα. Και πρέπει να υποστηρίξουμε επίσης και τους καταναλωτές, να δημιουργηθεί ένα κλίμα εμπιστοσύνης και να διασφαλίσουμε ένα πλαίσιο ασφάλειας για αυτούς. Έχουμε πολλά που πρέπει ακόμα να πράξουμε και έχουμε καθυστερήσει σε αυτό το θέμα οι, οι μπορούν να συνεισφέρουν σημαντικά. Άρχισα λέγοντας ότι έχω αισιοδοξία. Πιστεύω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε να προχωρήσουμε. Έτσι ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πιστεύω ότι πρώτα απ' όλα <clears throat> ότι έχουμε πολύ καλή βάση, θετικά θεμέλια με τα όσα συζητούμε για αυτή την έκθεση. Εγώ πιστεύω τρία ζητήματα είναι πολύ σημαντικά ως άξονες. Πρώτος άξονας, στην ψηφιακή οικονομία. Δεν υπάρχει καμιά ευκαιρία να είναι κανείς ο δεύτερος. Πρέπει πάντα να είναι ο πρώτος. Αυτό θα δρέψει τις δάφνες και τους καρπούς. Και αυτό πρέπει να ε, αλλάξει την οτροπία των ανθρώπων. Αν θα θέλει κάποιος να προσπαθήσει να υπερασπιστεί την Ευρώπη κρατώντας άλλους εκτός σε ένα στεγανό πλαίσιο, το αποτέλεσμα θα είναι ότι θα υποστηρίξουμε από τον ανταγωνισμό της δικές μας επιχειρήσεις. Αν θέλουμε να είμαστε ε, αποτελεσματικοί πρέπει να υπάρχει ένα ανοιχτό πλαίσιο και να είμαστε αποδοτικοί με καλές επιδόσεις σε ένα ανοιχτό πλαίσιο και για την ε, ροή των δεδομένων και για το πώς θα αντιμετωπιστούν τα θέματα του παγκόσμιου ανταγωνισμού από εμάς. Δεύτερος άξονας. Αν θέλουμε να είμαστε πρωτοπόροι και προπομπή, πρέπει να δεχθούμε τις αλλαγές που θα συνεπιφέρει η ψηφιοποίηση. Πρέπει να έχουμε ένα ανοιχτό πνεύμα, με ανοιχτή νοοτροπία να αντιμετωπίσουμε τις εξελίξεις και τα τεκτενόμενα ξέρουμε τα θέματα σε σχέση με αυτή την παγκοσμιοποίηση. Πρέπει αυτά να τα εξετάσουμε ως ευκαιρίες να μετατρέψουμε, να τροποποιήσουμε την οικονομία μας, να είμαστε πιο αποτελεσματικοί, με καλύτερες επιδόσεις. Και τέλος, τώρα σύντομα θα έχουμε την ψηφιοποίηση και στο διαδίκτυο, στο ίντερνετ αυτή θα είναι η χρονική στιγμή όπου οι επιχειρήσεις θα πρέπει να κάνουν ένα νέο βήμα προς τα εμπρός για να μετεξελιχθούν. Συζητώντας τα θέματα του διαδικτύου, το βλέπουμε αυτό. Το διαδίκτυο και η ψηφιοποίηση όχι μόνο θα επιβληθεί σε όλους τους τομείς, αλλά θα αλλάξει και την οτροπία και τη λογική, το πνεύμα στην κοινωνία μας. Για να είμαστε εμείς οι πρώτοι, οι πρωτοπόροι, πρέπει να έχουμε τις καλύτερες προϋποθέσεις από πλευράς υποδομών. Πρέπει να διασφαλίσουμε το ότι εμείς θα είμαστε οι πρωτοπόροι όσον αφορά το κινητό διαδίκτυο, για παράδειγμα, mobile internet, γιατί στις ε, υπηρεσίες, στις κινητές, ε, σε όλες ε, τις συναλλαγές που θα απορρέουν. Να είμαστε οι πρώτοι. Μπορούμε να το επιλέξουμε αυτό. Ή εμείς να είμαστε πρωτοπόροι ή θα είναι οι Αμερικανοί ή οι Ασιάτες. Πρέπει να δράσουμε ώστε οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να μπορούν στις τηλεπικοινωνίες και παντού να είναι οι πρωτοπόρες. Ευχαριστώ. Thank Σας ευχαριστώ οι συνεισηγήτρες και καλή τύχη σας εύχομαι. Δεν θα είναι καθόλου εύκολο αυτό το εγχείρημα για σας. Παρακολουθώ από την πλευρά από πολύ κοντά τα όσα συμβαίνουν και έχουμε <clears throat> αντιπρόεδρο που πραγματικά μπορεί να επιληφθεί αυτών των θεμάτων. Βλέποντας τις επιδόσεις για τον εξυγχρονισμό όσον αφορά τα θέματα αυτά από πλευρά του έχοντα θάρρο ε, και ε, καλές επιδόσεις θα στεφθεί με επιτυχία το εγχείρημα. Πρέπει να υποστηρίξουμε κάθε λέξη που λέει ο Αντιπρόεδρος ε, σε αυτή την επανάσταση, την ψηφιακή, χρειαζόμαστε πραγματικά να βοηθήσουμε κάποιον να βοηθήσει τους άλλους, εμάς δηλαδή, να προχωρήσουμε εμείς από πλευράς μας. Θα είναι δύσκολο το εγχείρημα διότι δεν είναι εύκολες λαϊκίστικες οι επιλογές. Αν ακολουθηθούν τέτοιες λαϊκίστικες επιλογές βραχυπρόθεσμα μόνο θα υπάρχουν κάποια ωφέλη τιμωρώντας επιχειρήσεις όπως συμβαίνει στην Uber για παράδειγμα στη Γαλλία με την Uber δεν είναι πράγματα τα οποία βοηθούν πλήττουμε το μέλλον της ψηφιοποίησης και το μέλλον της Ευρώπης σε αυτή την επανάσταση τιμωρώντας επιχειρήσεις. Και δεν υπάρχει προοπτική σε αυτό το εγχείρημα. Πρέπει να πάμε πιο βαθιά, σε μεγαλύτερη έκταση και βάθος. Και εδώ όταν βλέπουμε ότι υπάρχει κάποια αμερικανική, κάποια εταιρεία η οποία και δεν πρέπει να θεωρείται μόνος αμερικανική, πρέπει να λυθούν πολύ σκληρές αποφάσεις. Δεν είναι εύκολες οι επιλογές, Ας ρωτήσουμε, ας ζητήσουμε από τους επαΐοντες μια ισορροπημένη τέτοια προσέγγιση. Και έτσι μπορούμε να συνδράμουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προαγάγει αυτή την επιλογή και να έχουν επιλογές οι νέοι μας στην Ευρώπη για τις ζωές τους. Ευχαριστώ. Sorry that you're lost. Εσείς παρακαλώ έχετε τον λόγο. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Σε λίγα δευτερόλεπτα, πολύ σύντομα από πλευράς μου. Θα ήθελα να προσθέσω κάποια θέματα. Πρώτα, θα ήθελα να ευχαριστήσω τις συνεισηγήτριες διότι προετοίμασαν τα θεμέλια, τη βάση αυτή για το έργο που πρέπει να επιτελέσουμε. Σας ευχαριστούμε επίσης και για τη συζήτηση που διεξήχθη σήμερα. Ακούσαμε πολλές παρεμβάσεις που δείχνουν ότι βρισκόμαστε στην αφετηρία αυτών των πραγμάτων, αυτής της διαδικασίας. Δεν θέλω να ακουστούν λαϊκίστικες οι δικές μου αυτές παρεμβάσεις στα σχόλιά μου να πούμε ότι πρέπει να προστατευτούμε από κάποιους. Αλλά τρεις παρατηρήσεις θέλω να κάνω. Στα έγγραφα αυτά σήμερα μπορεί κανείς να δει κάτι. Να δει ότι πρέπει να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Υπάρχει αμερικανική εταιρεία με τεράστια με παραγωγή κομπιούτερ που ασχολούνται με τα μεγαδεδομένα, με τα με το υπολογιστικό και λοιπά. Υπάρχουν λοιπόν επιχειρήσεις ε, στην Ευρώπη που μπορούμε, μπορούν να συναγωνιστούν κάποιες επιχειρήσεις αμερικανικές και όχι μόνο. Αλλά δυστυχώς έχουν ε, και πολλές από τις επιχειρήσεις ε, στην Ευρώπη έχουν χαθεί, έχουν κλείσει. Η εταιρεία όπως η ξέρουμε ότι έκλεισε διότι έκανε λάθος με τα λειτουργικά της στη βιομηχανία των ΤΑΦΙΕ χάσαμε τον μάχη των λειτουργικών συστημάτων και χάνουμε σιγά σιγά και τη μάχη για τους μεγάλες πλατφόρμες του ίντερνετ. Και περνάμε σε ένα σύστημα πλατφόρμων κλειστών όχι, που δεν είναι ανοιχτέ στον ανταγωνισμό. Αυτό θα πρέπει να το εξετάσουμε. Ευχαριστώ πολύ, παρατηρή πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε ακόμα τέσσερα λεπτά διερμηνίας διότι μερικοί διερμηνείς θα χρειαστεί να αποχωρήσουν. Η Επιτροπή λοιπόν θα πρέπει να απαντήσει στα όσα υπόθηκαν τις τελευταίες ώρες. Ο κ. Γκράφ αρμόδιος για τη ψηφιακή οικονομία, θέλει να κάνει κάποιες παρατηρήσεις. Σίγουρα θα έχει την ευκαιρία να αντιδράσει σε κάποια άλλη στιγμή. Θα μιλήσω λίγο πιο γρήγορα, θα πω λίγο, κάπως λιγότερα πράγματα. Καταρχήν καλωσορίζουμε αυτή την έκθεση. Νομίζω πως οι προτεραιότητες ε, είναι ουσιαστικές, ε, όπως το επίπεδο φιλοδοξίας θα χρειάζεται να ανεληφθούν συγκεκριμένε δράσεις και να ε, προχωρήσουμε στην εφαρμογή. Είναι λοιπόν ευπρόσδεκτα όλα αυτά η έκθεση της Κομισιόν αν εγκριθεί τον Ιανουάριο θα μπορέσουμε να λάβουμε υπόψη την ε, έκθεση αυτή. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι έχουμε ε, μια κοινή ανάλυση των προβλημάτων. Συμφωνούμε ότι ένα από βασικά προβλήματα για την έλλειψη ενία ψηφιακή αγορά είναι αυτό του κατακαιρματισμού. Ελάχιστη εναρμόνιση ακολουθήθηκε τα τελευταία χρόνια και τελικά Έχουμε 38 τελικούς ε, ε, κανόνες και ρυθμίσεις. Ε, αναφέρθηκε ότι αν είστε μια μικρή επιχείρηση πρέπει να ασχοληθείτε με αυτό 28 φορές. Ως καταναλωτής δεν ξέρετε αν θα τύχετε ικανής προστασίας από τα διάφορα νομικά συστήματα. Χρειάζεται λοιπόν να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Επίσης άκουσα πολλές ε, ουσιαστικές αρχές που τόνισαν τα μέλη με ολιστική προσέγγιση. Δεν πρόκειται για ένα μενού από το οποίο διαλέγουμε. Πρέπει να δουλέψουμε ομού, να εργαστούμε για αρχές ε, των πρακτικών. Χρειάζεται να είμαστε τεχνολογικά ούτε διότι η τεχνολογία αλλάζει γρήγορα. Πρέπει να είμαστε υπέρ της ε, καινοτομίας να λάβουμε υπόψη μας ότι δεν είμαστε μόνοι αποτελούμε μέρος μιας ευρύτερης οικονομίας με το οποίο είμαστε πολύ στενά συνδεδεμένα. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι υπάρχει ένα ισότιμο επίπεδο ανταγωνισμού, ε, ότι υπάρχει ασφάλεια και δικαιοσύνη. Αναφέρθηκα σήμερα πολλέ αρχέ ε, με τι οποίε συμφωνεί η Κομισιόν. Ε, η Κομισιόν αναφέρθηκε ότι προσπαθεί να επιβάλλει στόχους στα κράτη-μέρη. Δεν είναι για αλήθεια κάτι τέτοιο. Εμεί δεν επιβάλλουμε στόχου, απλά μετράμε την πρόοδο. Δεν ε, θέτουμε στόχους. Εν συντομία τώρα, για μια σειρά συγκεκριμένων ζητημάτων, το ηλεκτρονικό εμπόριο, ίσως 25 πριν από 25 χρόνια. Ε, ξέραμε ε, ότι αυτό το εμπόριο το από ε, ιδιωτικέ επιχειρήσει. Τώρα θα πρέπει να περάσουμε ε, το, τα, τις περιορισμούς του geo-blocking. Και προς το παρόν δεν είδαμε να γίνεται αναφορά στην εκθέση σας. Φυσικά η αγορά χρειάζεται να παίξει το ρόλο της και πολύ, πολύ σωστά υπογράμμισαν τον ρόλο του δημοσίου τομέα, χρησιμοποιώντας ε, τα διαφορετικά ταμεία, βιομηχανία 0,4, πρόοδος θα πρέπει να επιτευχθεί, πρέπει να είμαστε ηγέτες ε, στην τεχνολογία 5G, πρέπει να υπάρχει νομική ασφάλεια και ό,τι την πρόσβαση δεδομένων, την, ε, ε, την αξιοπιστία των δεδομένων Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Thank you, Mr. De Ευχαριστώ, κύριε De Graaf. Υπάρχει κάποιο άλλο ομιλητή από πλευρά Κομισιόν, όχι. Μια σύντομη παρέμβαση των εισηγητέ. Θα συνεχίσουμε να έχουμε κάποιε γλώσσες ε, γερμανικά, γαλλικά, ιταλικά, ρουμανικά, ελληνικά. Ε, οι υπόλοιποι διαδμοί θα χρειαστεί να αναχωρήσουν. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ όλους όσοι σχολίασαν, θα είμαι ιδιαίτερα σύντομη. Κάτι το οποίο έθιξαν πολλοί από εσάς είναι οι πλατφόρμες και τα σχόλια σας έδειξαν ότι δεν μπορούμε να έχουμε το one size, one size fits all, να έχουμε μια πλατφόρμα που να ισχύει για όλες τις περιπτώσεις. Για κάποια από τα ζητήματα που, με τα οποία επικριθήκαμε ότι η προστασία δεδομένων και τα ψηφιακά προσόντα, ή δεξιότητες ε, δεν εθίγησαν επαρκώς. Έχουμε αυτή την κοινή έκθεση. Υπάρχουν διάφορες ε, επιτροπές που έχουν ποικίλε αρμοδιότητες και η προστασία δεδομένων ανήκει στη ΛΥΜΠΕ που θα συζητήσουν όλα αυτά τα ζητήματα εκτενώς. Γι' αυτό λοιπόν δεν θέλαμε να υπερβούμε τις αρμοδιότητές μας. Τώρα σε ό,τι φορά τις υποδομές συμφωνώ πως αν δεν έχουμε πρόσβαση στο διαδίκτυο δεν μπορούμε να μιλάμε για ενιαία ψηφιακή αγορά. Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι πως αυτοί οι κανονισμοί, οι κανόνες που είναι τεχνολογικά ουδέτεροι για να μπορούν να εφαρμοστούν στο γυναικές. Το θέμα της φορολόγησης Σίγουρα αυτή παρεμποδίζει την ε, ενιαία αγορά. Και ειδικά ο τρόπος με οποίο ε, γίνεται η διαχείριση των φόρων. Μπορεί να υπάρχουν διαφορετικές συντελεστές, αλλά να έχετε ε, δυνατότητες συμπλήρωσης των, των δηλώσεων σου. Τώρα, για τη συμφωνία συμφωνώ ότι είναι ζήτημα κλειδί. Δεν θέλουμε να επιδιορθώσουμε κάτι το οποίο έχει ήδη σπάσει. Τώρα, σχόλια σχετικά με το σφαιρικό διαδίκτυο. Όταν μιλάμε για ψηφιακή ενία αγορά στην Ευρώπη, τα σημαντικότερα εμπόδια είναι πως υπάρχουν 28 διαφορετικά καθεστώτα. Αυτό θα πρέπει να εξετάσουμε στην συγκεκριμένη έκθεση. Και για να κλείσω, θεωρώ ότι έχει σημασία να μην χάσουμε το στόχο μας. Μιλάμε για ενιαία ψηφιακή αγορά. Ε, υπηρεσίες και προϊόντα μπορούν να ε, διασχίζουν τα σύντομα. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Ευχαριστώ. Γεπάρτ. ευχαριστώ πολύ. Και εγώ θέλω κυρίως να ευχαριστήσω. Να ευχαριστήσω για τα πολλά σχόλια. Ένα εκ προημίου. Η εθνική πρωτοβουλία μόνη της δεν επαρκεί. Δεν είναι η σωστή πορεία αυτή. Να μην πιστεύει κανείς ότι ένα κράτος μπορεί να βρει τις σωστές απαντήσεις για αυτή την ψηφιακή πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Μόνο οι ευρωπαϊκές μπορεί να είναι οι απαντήσεις και έτσι μπορούν να βρεθούν οι λύσεις. Ένα τομέα είναι πολύ σημαντικό που αναφέρθηκε από επιμέρου ευρωβουλευτέ ε, και είναι το θέμα των επιπτώσεων στην καθημερινή ζωή των πολιτών μας. Και αυτό πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο των ανησυχιών μας και των μελημάτων μας. Η προστασία των καταναλωτών φυσικά πρώτα, τα δικαιώματα των χρηστών σε όλους τους τομείς, αλλά και οι όροι εργασίας, προϋποθέσεις και όροι εργασίας για τους πολίτες ασκήθηκαν επικρίσεις ότι η Uber λέει υπέστη επικρίσεις στη Γαλλία μπορώ να το κατανοήσω πολύ καλά αυτό η Uber έχει ανεξάρτητους εργαζόμενους οι οποίοι δεν είναι καν ασφαλισμένοι κοινωνικά και ανταγωνίζονται άλλες επιχειρήσεις που υπάρχουν ήδη κάποιες δηλαδή που είναι πιο ακριβές στην παροχή υπηρεσιών, γιατί ασφαλίζονται και οι οδηγοί ταξί σε αυτές τις εταιρείες. Τι θέλουμε λοιπόν για τους εργαζομένους, να εργάζονται ανασφάλιστοι, δηλαδή να είναι ένα μη κοινωνικό πλαίσιο που θα δημιουργήσουμε. Για αυτούς ή θα δημιουργηθεί ένα κοινωνικό πλαίσιο κοινωνικής ασφάλισης και πρέπει να δούμε ότι είναι οι καταναλωτές και χρήστες που μπορούν να υποστηρίξουν και την οικονομία με αυτόν τον τρόπο. Όλα αυτά είναι θέματα που συνολικά πρέπει να αντιμετωπιστούν. Προστασία καταναλωτών, προστασία δεδομένων, ουδετερότητα των δικτύων. Έχουν πολύ μεγάλη εμβέλεια και σπουδαιότητα όλα αυτά και από κοινού με τι άλλε κοινοβουλευτικέ επιτροπέ που είναι συναρμόδιε θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτά τα θέματα επιμερίζοντα τι αρμοδιότητε μεταξύ μα και το δικαίωμα δηλαδή των δημιουργών, των παραγωγών, δικαιώματα πνευματική ή διανοητική ιδιοκτησία και συγγενή δικαιώματα. Και ένα θέμα στο οποίο νομίζω ότι όλοι μεταξύ άλλων συμφωνούμε είναι το θέμα των πλατφορμών δεν υπάρχει μία και μόνη πλατφόρμα ή πλατφόρμα. Υπάρχουν πολυμορφίες ε, πλατφόρμων και δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει ένας ορισμός για αυτές τις πολυσχηδείς δραστηριότητες αυτών των πλατφορμών μεταξύ ψαχτηρίων, μηχανών αναζητήσεων, πλατφορμών αναζήτησης, ε, έρευνας, ε, κοινωνικών τέτοιων μέσων που από κοινού θέλουν να συνεργαστούν και να εργαστούν και δεν έχουν εμπορικό σκοπό, δηλαδή κερδοφορία ή κερδοσκοπία. Όλα αυτά είναι διαφορετικά θέματα που πρέπει διαφοροποιημένα να τα αντιμετωπίσουμε με τον σωστότερο τρόπο, εξετάζοντας το τι είναι το πιο ενδεδειγμένο πολύ προσεκτικά για όλα αυτά και έτσι θα έχουμε διαφορετικές διαδρομές και πορείες Προσβλέπω και χαίρομαι στη μελλοντική, για τη μελλοντική αυτή συνεργασία. Θα έχουμε περαιτέρω συζητήσεις και με σκιώδεις εισηγητέ και εισηγητέ των άλλων κοινοβουλευτικών επιτροπών. Είναι πραγματική ευχαρίστηση να συνεργαζόμαστε έτσι με αυτόν τον τρόπο για να προαγάγουμε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Thank you very much everyone, um, Σας ευχαριστώ πολύ όλους για τη σημερινή συνάντηση. Σας επενθυμίζω ότι η προθεσμία υποβολή τροπολογιών λύγει την Πέμπτη και η ψηφοφορία θα λάβει χώρα στις 14 Δεκεμβρίου, Δευτέρα βράδυ, στο Στρασβούργο. Είναι θετικό το ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα λάβει υπόψη τα αποτελέσματα αυτής της ψηφοφορίας εργασίας της και να σας υπενθυμίσουμε ότι εδώ πέρα είναι πολλά τα ζητήματα. Και σίγουρα η έκθεση θα είναι ιδιαίτερα εμπεριστατωμένη και εκτενής. Ευχαριστώ και τον ε, Γιαρζιμπούζεκ ε, που συμπροέδρευσε μαζί μου. Να δώσω τον ε, τελικό λόγο λοιπόν στον ίδιο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε για την πολύ καλή αυτή συνεργασία με όλους τους συναδέλφους αλλά και τους βοηθούς, τους συμβούλους και οι πολίτες βεβαίω μας παρακολούθησαν. Είναι πολύ καλό που κάναμε αυτή τη συζήτηση όλοι μαζί για την ενιαία ψηφιακή αγορά, για τα δικαιώματα του καταναλωτή. Νομίζω ότι ο καθένα μπορεί να κατανοήσει πραγματικά και οι πολίτε μα να παρακολουθήσουν από κοντά αυτή τη συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ. Και καλή επιτυχία για την επόμενη συνάντηση. Διακόπη το μικρόφωνο της Πρόεδρου στις 14 Δεκεμβρίου. Φαντάζομαι θα είναι μεγάλη ψηφοφορία. Να είστε έτοιμοι λοιπόν.